Welcome uh, uh, Καλώς ορίσατε όλοι. Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα το πρωί με την Ελληνίδα Υπουργό Απασχόλησης και θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό νομίζω επανειλημμένα. Ελπίζω να έχετε την κάρτα σας για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε. Θα ξεκινήσουμε με την προσωρινή συμφωνία για τις οργανικές διαπραγματεύσεις που επιβεβαιώθηκαν από το ΚΟΕΠΕ. Άρχεται η ψηφοφορία, ψηφίζεται. Ένας παραπάνω Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα παρακαλώ. Πέρα στις ψηφοφορίες 42 υπέρ και 8 κατά. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε. Α, πρόεδρε, Δεν ακούγεται η ισπανική διερμηνία, λέει η κυρία. Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια τεχνικά προβλήματα με τη διερμηνία. Από το πρωί συνήθως τα προβλήματα αυτά δημιουργούν μικρές καθυστερήσεις, αλλά δεν θα πρέπει νομίζω να ξεκινάμε εξ αρχής κάθε φορά. Συνεχίζουμε λοιπόν με την ε, γνωμοδότηση για το γενικό προϋπολογισμό, συμβιβαστική α, ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, δεκτή. Τροπολογία 1, έχει καταπέσει 2, 3 και 4 ναι. Συμβιβαστική β, υπέρ, κατά, δεκτή. Τροπολογία 7. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. 27 ψήφοι υπέρ, 2 κατά. Το 8 έχει καταπέσει. Συμβιβαστικό γάμα. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτών. 14. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβιβαστικό διαγλικό υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Συμβιβαστικό ή αγγλικό, στην ίδια σελίδα, ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, δεκτή. 23 στην σελίδα 4. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβιβαστική F αγγλικό υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκ... Από την αρχή παρακαλώ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 30. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. G υπέρ κατά αποχές δεκτή. 31 δεύτερο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Απορρίπτεται. 38. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 39. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 40. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 42 υπέρ. Υπέρ επαναλαμβάνω κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 42 ψηφίζεται. Πέρα της ψηφοφορίας 29 υπέρ δεκτή. 43 τώρα με προφορική τροπολόγηση υπέρ κατά αποχές δεκτή. Αυτό σημαίνει ότι ψηφίζουμε τώρα το σύνολο της τροπολογημένης πρότασης. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 41 υπέρ λοιπόν. Ευχαριστώ. Πηγαίνουμε τώρα στη δημοσιονομική διαδικασία και στον αντίστοιχο κατάλογο αν έχετε. 57-70 υπέρ κατά αποχές δεκτό 5771 71 υπέρ κατά αποχές δεκτό 57-72 υπέρ κατά αποχές δεκτό 57-73 υπέρ κατά αποχές δεκτή πρόταση 5775 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5776 υπέρ κατά απορρίπτεται αλλά θα υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος για το 5776 παρακαλώ άρχεται η ψηφοφορία Πέρα της ψηφοφορίας, οι σοσιαλιστές έχουν έναν επιπλέον. Έτσι κι αλλιώς απορρίπτεται. Περνάμε λοιπόν στην 5774. Έχει καταπέσει, όχι έχει καταπέσει. Ποιοι είναι υπέρ, ψηφίζουμε λοιπόν, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Λοιπόν, 5774 ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία, πέρας της ψηφοφορίας. Έγινε δεκτή, 28 υπέρ, 23 κατά. 5777 τώρα, ποιοι είναι υπέρ Ποιοι είναι κατά. Δεκτή. 57-78 καταπίπτει. Περνάμε στην 57-79. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβιβαστική α υπέρ κατά αποχές δεκτή. 5781 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5782 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ για την 82 5782 άρχεται η ψηφοφορία πέραστη ψηφοφορίας απερίφθη 5785 υπέρ κατά αποχές απερίφη 5786 υπέρ κατά δεν ψηφίζουν οι σοσιαλιστές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 5786 άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Απερίφθη. 57-84. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 57-73. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 57-87, 89 συγγνώμη, κατά έγινε δεκτή, 88 υπερκατά υπέρ κατά αποχές απερίφη, 57-87 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η επόμενη καταπίπτη Πηγαίνουμε στην 57-95 υπέρ υπέρ, κατά, αποχές, απερίφη. 57-96 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφη. 57-94 υπέρ, κατά, αποχές, Απερίφη. Συμβιβαστική β, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 58.00 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 57.99 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή 58.01 υπέρ κατά αποχές δεκτή 58.02 υπέρ κατά απερίφθη 5803 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 5804 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτός, δεκτή, συγγνώμη. 5805 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφη. 5805 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 5807 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 5808 υπέρ κατά αποχές απερίφη. 5810 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 5811 υπέρ κατά αποχές δεκτή 58-12 υπέρ κατά αποχές απορρίφθη θα ελέγξουμε τώρα την 58-12 ψηφίζεται τέλος της ψηφοφορίας γίνεται δεκτή η 58-12 58-13 τώρα, υπέρ. Α, την 58-14 τότε πρέπει να ψηφίσουμε λέει η πρόεδρος, αλλά διακόπτει. Θα ψηφίσουμε την 58-13. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 58-14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 58-15 Την 14 την ψηφίσαμε λέει η Πρόεδρος. Έλεγχος τότε άρχεται η ψηφοφορία για τη 14. Τέλος της ψηφοφορίας. Είχε γίνει πράγματι δεκτή διορθώνει πρόεδρος. 58-15. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Δεκτή. 58-16. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 58-17. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 58-18 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 58-19 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 58-20 υπέρ, κατά, αποχές θα έλεγα δεκτή, αλλά μιας και έκανα λάθος προηγουμένως θα ζητήσω να υπάρξει έλεγχος για την 58-20. Ψηφίζετε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. Απερίφθη. 58-21. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 58-22 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 58-23 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 58-24 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 58-25 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 58-27 ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, αποχές απεριφθεί. ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 58-26 ψηφίζεται. Τέλος. Απερίφθη. 58-26. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 58-30. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Ηλεκτρονικός έλεγχος λοιπόν για την 58.30 30 Ψηφίζεται. Τέλος. Απερίφθη. 58-31. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απερίφθη. 58-29. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα έλεγα ότι γίνεται δεκτή, αλλά θα την ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζεται την 58-29. Πέρα τη ψηφοφορία. Έγινε δεκτή. 58-32. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 58-33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. ηλεκτρονικός έλεγχος της 5833. Ψηφίζεται. Τέλος. Απερίφη. 5834. οκτώ τριάντα τέσσερα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 58-35 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 58-36 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος. Τέλος. Απερίφθη. Ε, ε, Θέλω να σας ενημερώσω ότι ο κύριος Φερχόφστατ θα έρθει νωρίτερα από ό,τι προβλέπετε στο πρόγραμμά μας. Θα είναι εδώ στις 4 παρα 20. Θέλει να αρχίσουμε νωρίτερα. Αυτό βέβαια είναι καλύτερο και για μας. Θα είναι εδώ λοιπόν σε 10 λεπτά από τώρα. Οπότε πολύ μικρή διακοπή, διάλειμμα, σε 10 λεπτά όμως θα είναι εδώ. Friends, we start a uh, uh, bit earlier because uh, Mr. Verhofstadt is already here, and it's good so that we proceed with our meeting. Α, ε, μπορούμε να αρχίσουμε λίγο νωρίτερα. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Φερχόφστατ και μετά θα μπορέσουμε να υποβάλουμε ερωτήσεις και να συζητήσουμε και μαζί του. Λοιπόν, κύριε Φερχόφστατ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Και πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Ευχαριστώ και σας την Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής αυτής για την συμβολή τους τις τελευταίες εβδομάδες και τους τελευταίους μήνες στο ψήφισμα που ετοίμασε το Κοινοβούλιο, που ψήφισε, αλλά και στις ερωτήσεις και συζητήσεις για τα δικαιώματα των πολιτών που συζητούμε επί του παρόντος. Επιτρέψτε μου λοιπόν να προχωρήσω σε μια σύντομη εισαγωγή αναφερόμενος σε δύο ζητήματα κύρια. Πρώτον, θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω πώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμπλέκεται επί του παρόντος στις ε, τρέχουσες διαπραγματεύσεις. Δεύτερον, θα προσπαθήσουμε να δούμε μαζί πού έχουμε φτάσει. Αυτό θα είναι σύντομο βέβαια, πολύ σύντομο στην παρέμβασή μου. Και στη συνέχεια θα μιλήσω λίγο για το πώς σκεφτόμαστε να προχωρήσουμε τις επόμενες εβδομάδες. Τι συζητάμε αυτή την εβδομάδα, σε αυτό το γύρο των διαπραγματεύσεων και ποιος θα είναι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τις επόμενες εβδομάδες. Όσον αφορά λοιπόν την ε, οργάνωση, το οργανωτικό τμήμα των διαπραγματεύσεων αυτών. Γνωρίζετε ότι και εμείς και το Συμβούλιο έχουμε ορίσει τον Μισελ Μπαρνιέ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαπραγματευτεί από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό σημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει δημιουργήσει μια ομάδα εργασίας Brexit και εμείς έχουμε δημιουργήσει μια steering committee. Αυτοί έχουν ομάδα εργασίας, εμείς έχουμε διευθυντική επιτροπή εμείς. Έχει σημασία αυτό σημειολογικά το ότι η λέξη χρησιμοποιεί ο καθένας ομάδα εργασίας λοιπόν στο Συμβούλιο που σημαίνει ότι βασίζεται σε εκπροσώπους των 27 χωρών μελών της Ένωσης, ενώ η ομάδα steering, η διευθυντική ομάδα κατά κάποιο τρόπο, δουλεύει υπό την διάσκεψη των Προέδρων και η ομάδα αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελείται από εκπροσώπους των ε, ομάδων που στήριξαν το πρώτο ψήφισμα για το Brexit που εγκρίθηκε πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές από την Ολομέλεια. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν προχωράμε και αυτή η ομάδα η steering συνεδριάζει κάθε εβδομάδα περίπου και έχει συνεχείς επαφές με τον Μισελ Μπαρνιέ και ο Μισελ Μπαρνιέ κάθε εβδομάδα και αυτός παρουσιάζει τα πράγματα. Πώς δηλαδή θα προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις, ποια θα είναι η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε τη Δευτέρα θα βρεθώ πάλι μαζί του με την ομάδα αυτή steering και θα ακούσουμε και για τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων γιατί οι διαπραγματεύσεις αυτές όπως ε, ξέρετε ακολουθούν έναν κύκλο τεσσάρων εβδομάδων. Ετοιμάζουμε τις θέσεις μας, οι δύο πλευρές την πρώτη εβδομάδα, τη δεύτερη εβδομάδα ανταλλάσσουμε τι απόψει μα. στη δεύτερη εβδομάδα που είναι αυτή γίνονται οι διαπραγματεύσει αυτές κάθε αυτές. Εκεί βρισκόμαστε τώρα και τέταρτη εβδομάδα, η επόμενη, γίνεται το debriefing. Δηλαδή υπάρχει η ενημέρωση στο Ενωμένο Βασίλειο από τους δικούς τους και από τον Μπαρνιέ σε εμά στις δύο αυτές ομάδες του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσημα λοιπόν, όπως είπαμε, βρισκόμαστε στην τρίτη εβδομάδα των διαπραγματεύσεων. 19 Ιουνίου ξεκίνησε ο πρώτος γύρος, 20 Ιουλίου ξεκίνησε ο δεύτερος γύρος και ο τρίτος γύρος ξεκίνησε την ε, Δευτέρα. Ο πρώτος γύρος διαπραγματεύσεων ήταν η εκκίνηση των διαπραγματεύσεων ουσιαστικά. Ο δεύτερος γύρος που άρχισε 20 Ιουλίου ήταν η παρουσίαση των θέσεων των δύο πλευρών. Και ο τρίτος γύρος που άρχισε τη Δευτέρα είναι η διασαφήνιση. Ελπίζω κάποια στιγμή να φτάσουμε και σε διαπραγματεύσεις, σε ένα γύρο διαπραγματεύσεων, πραγματικών διαπραγματεύσεων. Έχουν δημιουργηθεί τρεις ομάδες μέσα στην διαπραγμάτευση. Σε αυτούς τους πρώτο, δεύτερο και τρίτο γύρο. Μία αφορά τα δικαιώματα των πολιτών. Και όπως ξέρετε είναι στοιχείο κλειδί για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θέλουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα να σταματήσει αυτή η βεβαιότητα που δημιουργήθηκε από το Brexit όσον αφορά τους πολίτες, τους Ευρωπαίους που ζουν στον Ηνωμένο Βασίλειο και τους Βρετανούς που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και για να μην υπάρχει αυτή η βεβαιότητα πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία για τα δικαιώματά τους. Υπάρχει και μια δεύτερη ομάδα εργασίας στις διαπραγματεύσεις λοιπόν που δημιουργήθηκε και έχει να κάνει με τους ε, χρηματοοικονομικούς διακανονισμούς Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ξέρετε, παρουσίασε ένα λεπτομερές έγγραφο για το ποιος θα πρέπει να είναι αυτός ο οικονομικός διακανονισμός. Και η τρίτη ομάδα εργασίας που δημιουργήθηκε είναι για άλλα θέματα. Υπάρχει ένας ολόκληρος κατάλογος πιο συγκεκριμένων ζητημάτων που θα πρέπει να εξεταστούν πριν αποσυρθεί το ΕΒ το 2019. Το πιο γνωστό είναι η Ευρατόμ και η πυρηνική ασφάλεια. Συνολικά υπάρχουν κάπου 7 θέματα τα οποία περιλαμβάνονται σε αρμοδιότητες της τρίτης ομάδας εργασίας. Και αποφασίσαμε να μην έχουμε μεν ομάδα εργασίας, αλλά να υπάρχει διάλογος ανάμεσα στους αναπληρωτές και από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον κύριο Ρόμπινς που είναι υπεύθυνο για τον Brexit στον Ηνωμένο Βασίλειο. Για το θέμα της Ιρλανδίας και των συνόρων ανάμεσα στη Βόρεια Ιρλανδία και τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Υπάρχουν ε, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο τέσσερις διαφορετικές ε, ομάδες, τρεις επίσημα ομάδες εργασίας όπως τις λέμε, δικαιώματα των ε, πολιτών, οικονομικά ζητήματα και άλλα θέματα διαχωρισμού και το τέταρτο είναι ο διάλογος, όπως σας είπα, μεταξύ των δύο αναπληρωτών για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα σύνορα ανάμεσα στην Ιρλανδική Δημοκρατία και τη Βόρεια Ιρλανδία. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Πώς οργανώνονται αυτές. Και σας υπενθυμίσω ότι βρισκόμαστε στον τρίτο γύρο διαπραγματεύσεων. Ο τέταρτος προβλέπεται για τα τέλη Σεπτεμβρίου. Και τότε θα αρχίσει και ένα άλλο όταν ολοκληρωθεί αυτός και αυτός ο πέμπτος θα είναι τον Οκτώβριο. Τώρα για την ουσία των διαπραγματεύσεων. Είμαι στο δεύτερο σημείο μου δηλαδή. Εδώ βέβαια είναι γνωστά, έτσι. Σπρώχνουν ανοιχτέ πόρτες όπως λέμε εμείς στο Ολλανδικά λέει ο κύριος Φερχόστατ. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σας πω ότι υπάρχει αργή πρόοδος. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι και από τις δύο πλευρές χρειαζόμαστε τις τοποθετήσεις για κάθε ζήτημα χωριστά. Γιατί αν σε πραγματεύσεις έρχεται μόνο η μία πλευρά με τη δικιά της τοποθέτηση, η ε, άλλη δεν αντιδρά, οπότε έτσι δεν μπορούν να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Όμως συγχρόνω πιστεύω ότι αυτό το οποίο είναι ξεκάθαρο είναι ότι όλοι πιστεύουμε, και δύο πλευρές δηλαδή, ότι δεν είναι καθόλου καλό να προχωράμε χωρίς συμφωνία. Δηλαδή αν το αποτέλεσμα είναι έλλειψη συμφωνίας, αυτό είναι κακό για όλους και για τις δύο πλευρές. Άρα δεν αποτελεί επιλογή να προχωρήσουμε έχοντας το μυαλό μας ότι δεν θα καταλήξουμε. Έπειτα, από πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου υπάρχει καλύτερη κατανόηση όσον αφορά τη μεταβατική περίοδο. Ξέρετε ότι υπήρξε θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την πρώτη μέρα και θα το βρείτε και στο ψήφισμα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο. Από την αρχή εμείς είπαμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση 14-15 μήνες να συμφωνήσουμε για απόσυρση συμφωνία δηλαδή που να περιλαμβάνει και τις οικονομικές διευθετήσεις και τα ελληνικά σύνορα και τα δικαιώματα των πολιτών και όλα τα υπόλοιπα και επιπλέον σε λεπτομέρειες να έχουμε και συμφωνία για τις μελλοντικέ σχέσεις μεταξύ μας. Για να γίνει αυτό, μέσα σε 14 μήνες, για μας από την αρχή αυτό ήταν αδιανόητο. Γι' αυτό και το ψήφισμα το οποίο εγκρίνατε κι εσείς περιλαμβάνει μία παράγραφο η οποία αναφέρεται σε μία μεταβατική περίοδο η οποία θα είναι περιορισμένη στο χρόνο. Είπαμε τρία χρόνια για παράδειγμα, θα το θυμόσαστε έτσι. Οπότε τώρα αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο η αναγκαιότητα για μια τέτοια μεταβατική περίοδο. Το τι θα περιλαμβάνει αυτή η μεταβατική περίοδος, αυτό μένει να συζητηθεί βέβαια ακόμα. Πάντως όσο περισσότερο χρόνο χάνουμε τους επόμενους μήνες, τόσο πιο σαφές γίνεται ότι η μεταβατική αυτή περίοδος θα είναι η παράταση της σημερινής κατάστασης, του status quo δηλαδή. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να φανταστούμε σε λίγες εβδομάδες ή μήνες να έχουμε καταλήξει σε ένα νέο σύστημα. Πάντως, είπαμε, η συμφωνία είναι κάτι καλύτερο από την έλλειψη συμφωνίας. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, θα χρειαστούμε μία μεταβατική περίοδο. Θα χρειαστούμε το χρόνο αυτό της μεταβατικής περίοδου για να αποφασίσουμε ποια θα είναι η μελλοντική σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ηνωμένο Βασίλειο. Και η αρχή αυτή γίνεται όλο και περισσότερο αποδεκτή από όλους της μεταβατικής περίοδου. Και όπως θα έχετε διαπιστώσει κι εσείς, το Ηνωμένο Βασίλειο τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχει προβεί και σε διάφορες ανακοινώσεις, κάποιες είναι τοποθετήσεις, ε, κάποιες άλλες είναι τοποθετήσεις εταιρική σχέσης και τέσσερις από τις εφτά αυτές αφορούν τις μελλοντικέ σχέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ βέβαια δεν ήρθα να σχολιάσω από αυτόν και γιατί όχι, γιατί άποψή μας είναι ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο στη συμφωνία απόσυρσης του Ηνωμένου Βασιλείου πριν πούμε στις συζητήσεις για τις μελλοντικέ μας σχέσεις και δεν πιστεύουμε ότι έχουμε προχωρήσει αρκετά όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου για να μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο. Δεν έχουμε προχωρήσει αρκετά στα τρία δηλαδή κεφάλαια που σας είπα για να μπούμε στο κεφάλαιο των μελλοντικών σχέσεων. Δεν σημαίνει ότι βέβαια πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία αποχώρησης, ε, συμφωνήσαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι εφόσον έχει υπάρξει επαρκής πρόοδος, τότε μπορούμε να αρχίσουμε να συζητάμε για τις μελλοντικέ μας σχέσεις. Όμως, σίγουρα θα σημειώσατε ότι αυτά τα έγγραφα τα οποία παρουσιάστηκαν από τον Ηνωμένο Βασίλειο για τις μελλοντικέ σχέσεις ξεκινούν από την ιδέα που λέει ότι δεν θα είναι αρμόδιο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για αρμοδιότητες που έχουν να κάνουν εξωτερικό εμπόριο. Και δεν θα υπάρχει και συνέχεια πληρωμών προς τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έρχομαι Τώρα, στο θέμα των δικαιωμάτων των πολιτών, γιατί ξέρω ότι η δικιά σας ε, η Επιτροπή εμπλέκεται σε αυτές τις συζητήσεις και θέλω να έρθω στα ζητήματα της ε, συνθήκης που έχουν να κάνουν με την απόσπαση των εργαζομένων, με τον συντονισμό των συστημάτων ασφάλειας. Αυτά είναι στοιχεία κλειδί για τα δικαιώματα των πολιτών. Γενικά μιλώντας πρώτα. Και οι δύο πλευρές κατέληξαν σε έναν πίνακα δημοσιοποιείται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Ηνωμένο Βασίλειο, την κυβέρνησή του. Ένα πίνακα λοιπόν συγκριτικό ανάμεσα στις θέσεις. Και με πράσινο χρώμα είναι ε, τα σημεία στα οποία συμφωνούμε, κόκκινο είναι τα σημεία όπου δεν συμφωνούμε και κίτρινο είναι το χρώμα που δηλώνει ότι χρειάζεται περισσότερη δουλειά και περισσότερες διευκρινήσεις. Οπότε αποκλήσεις υπάρχουν για διάφορα ζητήματα. Υπάρχει συζήτηση για την επανένωση οικογενειών, για παράδειγμα, μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Υπάρχει το θέμα του επιπλέον διοικητικού βάρους η έλλειψη αναγνώρισης των εισφορών στην κοινωνική ασφάλιση μετά την αποχώρηση. Και θα επανέλθω. Δεν υπάρχει ε, αρκετή σαφήνη για τα δικαιώματα των εργαζομένων και για άλλα θέματα που έχουν να κάνουν ε, με τα δικαιώματα ε, του εκλέγην και κάποια άλλα οικονομικά δικαιώματα ή επαγγελματικά. Αυτά τα δύο τελευταία έχουν μπει με κίτρινο χρώμα. Άρα χρειάζονται παραπάνω συζήτηση και διευκρινήσεις. Συνεπώς, εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε με την διάσκεψη των Προέδρων στην Διευθυντική Ομάδα είναι να πιέσουμε στις διαπραγματεύσεις και τις δύο πλευρές να προχωρήσουν περισσότερο και να καταλήξουν όσον αφορά τα δικαιώματα των πολιτών. Γιατί δεν μπορούμε να διανοηθούμε 14-15 μήνες αβεβαιότητα για τους πολίτες. Και να ξέρετε ότι έχω φτάσει σε μένα εκατοντάδες επιστολών, χιλιάδες τώρα θα έλεγα, από ανθρώπους οι οποίοι έρχονται σε επαφή με το Κοινοβούλιο και λένε «Μα κοιτάξτε, εμείς δεν ξέρουμε ποιο είναι το καθεστώς μας» και δίνουν και συγκεκριμένα παραδείγματα και ρωτάνε τι πρέπει να κάνουμε. Και δεν έχουν να κάνουν μόνο με Ευρωπαίους που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και με Βρετανούς που ζουν σε κάποια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό που επίσης βλέπουμε, και είναι το πιο τρομερό παράδειγμα, ήταν μια επιστολή που εστάλει από το Υπουργείο Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου σε εκατοντάδε Ευρωπαίου πολίτες που τους έλεγε ότι πρέπει να εγκαταλείψουν το Ηνωμένο Βασίλειο. Εντάξει, αργότερα. Μετά είπαν ότι ήταν λάθος η επιστολή αυτή. Αλλά η αίσθηση που δημιουργείται, όπως καταλαβαίνετε, όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ότι γίνεται μια προσπάθεια να εκλειφθούν οι Βρετανοί στην Ευρώπη σαν ξένοι και οι Ευρωπαίοι στο Ηνωμένο Βασίλειο σαν ξένοι. Προς το παρόν ισχύει βέβαια η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Μέχρι τη στιγμή της αποχώρησης πρόκειται για Ευρωπαίους πολίτες. Οι Ευρωπαίοι και οι Βρετανοί είναι όλοι Ευρωπαίοι πολίτες και πρέπει να τυχαίνουν της ίδιας μεταχείρισης βάσει των ευρωπαϊκών κανόνων και όχι αλλιώς. Αλλά όλο και περισσότερο βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες δικητικές πρακτικές που αρχίζουν να εφαρμόζονται, που πιέζουν τους Ευρωπαίους στον Ηνωμένο Βασίλειο να πάνε και να ζητήσουν ε, ειδικά έγγραφα και τούμπαλοι. Και γι' αυτό και οι πολίτες μας γράφουν και διαμαρτύρονται. Εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είμαστε εδώ για να πούμε ότι εμεί υποστηρίζουμε μόνο τη μία κατηγορία πολιτών και όχι την άλλη. Όχι. Όλους τους υποστηρίζουμε. Και τους Ευρωπαίους στο Ηνωμένο Βασίλειο και τους Βρετανούς που ζουν στην υπηρετική Ευρώπη. Και έρχομαι στο τρίτο μου σημείο. Τι κάνουμε αυτή τη βδομάδα. Αυτή τη βδομάδα στις διαπραγματεύσεις εξετάζουμε τρία κεφάλαια, τρία θέματα σε αυτόν τον τρίτο γύρο. Το πρώτο έχει να κάνει με τα δικαιώματα των πολιτών, κάτι που αφορά μέσα τη δικιά σας επιτροπή. Ε, θα επικεντρωθούμε στα θέματα κοινωνικής ασφάλισης και συντονισμού. Επίσης, για τα ζωρευμένα δικαιώματα, Θα δούμε μετά την αποχώρηση. Θα υπάρξει διαφορετική μεταχείριση ή οι πολίτες θα μπορούν και μετά την αποχώρηση να συνεχίζουν να συσσωρεύουν τα δικαιώματά τους. Αυτό είναι ένα στοιχείο κλειδί που πρέπει να λύσουμε. Έπειτα, οι διασυνοριακοί οι εργαζόμενοι. Στο έγγραφο των ΗΠΑ Βασιλείου δεν αναφερόταν καθόλου το πρόβλημα αυτό. Και το τρίτο που θα συζητηθεί είναι η αμοιβαία αναγνώριση δεξιοτήτων στο μέλλον, προσόντων, επαγγελματικών προσόντων. Επίσης θα συζητήσουμε περισσότερο για τους οικονομικούς διακανονισμούς. Αυτό δηλαδή που αναμένουμε από πλευράς του Ηνωμένου Βασιλείου είναι την αντίδρασή τους όσον αφορά το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του κ. Μπαρνιέ για τους οικονομικούς διακανονισμούς και το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να αντιδράσει σε κάτι που είναι προφανές για μένα, ότι δηλαδή αν υπάρχουν διάφορες νομικές υποχρεώσεις, αυτές οι νομικές υποχρεώσεις δημιουργούν στη συνέχεια και οικονομικές υποχρεώσεις που πρέπει να τηρηθούν, να ληφθούν υπόψη κλπ. Και το τρίτο έχει να κάνει με την Ιρλανδία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η πρώτη σας ζήτηση σε βάθος για τα θέματα της ε, περιοχής των συνόρων ανάμεσα στην Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία ε, θα ακολουθήσει. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει κυκλοφορήσει ένα μνημόνιο ιδιαίτερα αναλυτικό για το πώς βλέπει την εξέλιξη της διαχείρισης των συνόρων στο μέλλον και την συνεργασία της Βόρειας Ιρλανδίας ε, με την υπόλοιπη Ιρλανδία μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση εμπλέκεται σε πάρα πολλά προγράμματα στη Βόρεια Ιρλανδία. Δεν περιμένουμε εμείς να υπάρξουν ριζικές λύσεις σε όλα αυτά τα θέματα, περιμένουμε όμως και στο θέμα της οικονομικής διαφοράς και στο θέμα της αντιμετώπισης των προβλημάτων των πολιτών και στο πρόβλημα το Ιρλανδικό να υπάρξουν κάποια πρώτα μικρά βήματα. Τώρα εμείς σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρόθεση δική μου και της ε, steering group της αρμόδιας και της διάσκεψης των προέδρων την επόμενη εβδομάδα ελπίζω είναι να επανέλθουμε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με μία πρόταση ψηφίσματος για τα δικαιώματα των πολιτών. Νομίζω ότι έχει φτάσει η στιγμή που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με βάση το αρχικό ψήφισμα να μπορεί να διευκρινίσει το τι μπορεί να δεχτεί και τι δεν μπορεί να δεχτεί από την πρόταση η οποία έχει γίνει από πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου. Όπως γνωρίζετε η πρόταση του Ηνωμένου Βασιλείου ονομάζεται διακανονισμένο καθεστώς, settled status για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πετύσει ε, ατομικές αιτήσει από κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αποκτήσει το καθεστώς αυτό. Είναι κάτι το οποίο θεωρητικά θα πρέπει να γίνει χωρίς προβλήματα, χωρίς εμπόδιο, ενώ θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι γιατί να μην συνεχίσουμε την υπάρχουσα ουσιαστικά κατάσταση. Να δώσουμε εγγυήσει για τα δικαιώματα των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου που ζουν στην Ευρωπαϊκή Υπηρετική Ένωση και ταυτόχρονα να δοθούν εγγυήσεις για τους πολίτες της Ένωσης που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Γιατί πρέπει να δημιουργήσουμε ένα νέο καθεστώς το οποίο να δημιουργήσει μια νέα κατηγορία πληθυσμού στο σύστημα μετανάστευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τώρα, ο έλεγχος του συστήματος αυτού είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνεται μιας και αφορά σε πολίτες της Ένωσης από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εκεί τα επιχειρήματά μας είναι σαφή. Κανένας δεν αμφιβάλλει για την ποιότητα των δικαστηρίων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Αλλά είναι κάτι που πρέπει να διευκρινιστεί. Νομίζω λοιπόν ότι είναι και πλέον η ώρα. Πρόθεσή μου είναι να πάω στην Ολομέλεια στις 3 Οκτωβρίου την πρώτη ολομέλεια του μηνός ε, Οκτωβρίου, ημέρα Τρίτη, με ένα ξεκάθαρο ψήφισμα, το οποίο να λέγει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από εβδομάδες και μήνες συζητήσεων και διαπραγματεύσεων, λέγει το τι δέχεται και τι δεν δέχεται. Καλύτερα να το διευκρινίσουμε τώρα παρά στο τέλος του κύκλου διαπραγματεύσεων το 2019. Να διευκρινίσουμε λοιπόν τι είναι δυνατόν για μας, τι δεν είναι δυνατόν για μας και να επιβεβαιώσουμε τους στόχους μας. Στόχος μας βασικός είναι η προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών. Στόχος της δημοκρατίας, στόχος της ευρωπαϊκής δημοκρατίας δεν μπορεί να είναι η μείωση των δικαιωμάτων, αλλά αν μη τι άλλο η προστασία του ισχύοντος σημερινού επίπεδου και αναφέρομαι εδώ όχι μόνο στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ τους. Είναι πολίτες που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να προστατευτούν. Αυτή λοιπόν είναι η βασική φιλοσοφία της συγκεκριμένη πρότασης η οποία φυσικά θα είναι λεπτομερέστατη γύρω από την πρόοδο των διαπραγματεύσεων, ανάλογα με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Είναι απαραίτητο στο ψήφισμα αυτό επίσης να γίνουν αναφορές για τη Βόρεια Ιρλανδία και τη συνοριακή περιοχή. Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να αντιδράσει σε ένα αναλυτικό μνημόνιο το οποίο έχει προετοιμάσει η Βρετανική πλευρά για τον τρόπο διαχείρισης της μεθορίου ανάμεσα στην Ιρλανδική Δημοκρατία και τη Βόρεια Ιρλανδία. Εμείς είπαμε ότι δεν μας αρέσει η ιδέα των συνόρων, δεν θέλουμε να αποκατασταθούν, να σκληρύνουν τα σύνορα. Το λεγόμενο σκληρό σύνορο, hard border, το αποκλείουμε. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το διευκρινίζουμε. Και τέλος, αυτό θα είναι ένα επιπλέον μέσο για να μπορέσουμε να αναφερθούμε και στην συνολική πρόοδο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης. Είναι επαρκής η πρόοδος. Ναι ή όχι. Αν τα πράγματα πηγαίνουν πάρα πολύ αργά, όπως φαίνεται να πηγαίνουν τώρα, θα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο να επιβεβαιώσουμε ε, ότι η πρόοδος ε, είναι σαφής. Όλα αυτά λοιπόν Το θέμα λοιπόν των δικαιωμάτων των πολιτών, το θέμα το μεθοριακό, το θέμα της πρόοδου των διαπραγματεύσεων. Νομίζω ότι για ένα δημοκρατικό εκλεγμένο σώμα, δημοκρατικά εκλεγμένο σώμα όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι η στιγμή να κάνει μια πρώτη αξιολόγηση και μην αναμένει να έρθει το τέλος της χρονιάς. Και νομίζω ότι περισσότερες από τις ομάδες που εργάζονται στο εσωτερικό του steering group θα συμφωνήσουν με τις προτάσεις αυτές και έτσι θα μπορέσουμε να διευρύνουμε τον αριθμό των ομάδων που εργάζονται εκεί στο μέλλον και αυτό είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί. Λοιπόν, αυτή δεν ήταν μια σύντομη παρουσίαση αλλά δεν ήταν και ιδιαίτερα μεγάλη για το που βρισκόμαστε σήμερα. Είμαι στη διάθεση της Επιτροπής σας και μπορώ να επανέλθω αν θέλετε όταν έχουμε προχωρήσει λίγο περισσότερο. Σας ευχαριστώ. Δεν ήταν μια σύντομη παρουσίαση, είχε όμως νόημα. Είναι μια καλή εισαγωγή για μας που δεν παρακολουθούμε τις διαπραγματεύσεις από πάρα πολύ κοντά και σε λεπτομέρεια. είναι η δυνατότητα θα έλεγα να μπορέσουμε να θέσουμε ερωτήσεις. Θα δώσω το λόγο στους συντονιστές της Επιτροπής και όσοι το επιθυμούν μπορούν να ζητήσουν το λόγο. Ο Τόμας Μαν, Κλούνε, Θα προσπαθήσουμε να είμαστε πάρα πολύ αποδοτικοί στη συζήτηση γιατί ο κύριο Φερχόφστατ δεν μπορεί να μείνει. Θα αρχίσουμε λοιπόν με τους συντονιστές από το ΕΛΚ. Ο κύριος Κάσης έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Φερχόστατ που ήρθε εδώ να μας παρουσιάσει την κατάσταση. Δεν ξέρω αν έχει σημειωθεί αρκετή πρόοδο σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών, διότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ μία από τις ομάδες που αναφέρατε. Για τα δικαιώματα λοιπόν των πολιτών σε ό,τι αφορά τις ασφαλιστικές δικλείδες για τα δικαιώματα που έχουν αποκτήσει οι πολίτες που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, η ερώτησή μου έχει ως εξή. Τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε αυτοί οι άνθρωποι να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, για παράδειγμα, και στην ιατροφαρμακευτική ε, περίθαλψη. Έχετε κάποια πρόθεση να απαντήσετε σε αυτό, ε, υπάρχει ε, πράσινη επισήμανση, κόκκινη, κίτρινη, σύμφωνα με αυτήν την ε, ταξινόμηση που μας είπατε πριν. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε τώρα στους ε, σοσιαλδημοκράτες. Ε, ο κύριος Κουτιέρες έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ πολύ κύριε Φερχόστα για την παρουσίασή σας και για το γεγονός ότι ήρθατε εδώ στην Επιτροπή μας. Διότι βλέπετε πιστεύω πως είναι ζωτική σημασία να συντονιζόμαστε για αυτό το θέμα, γιατί είναι ένα πεδίο μάχης. Κακά τα ψέματα. Η Βρετανική κυβέρνηση, που αποδυναμώθηκε βέβαια μετά από τις τελευταίες εκλογές που οργάνωσε η κυρία Μέη, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η ενιαία αγορά, η εσωτερική αγορά. Και το μόνο που θέλουν είναι να έχουν δικαιώματα σε αυτήν. Βέβαια έχει τεθεί και το θέμα των δικαιωμάτων των πολιτών και χαίρομαι που μας είπατε ότι φαίνεται να υπάρχει ενδιαφέρον και από τις δύο πλευρές γι' αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματα των πολιτών πάνε χέρι-χέρι με το δικαίωμα πρόσβαση στην εσωτερική αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου μετά την αποχώρηση. Πάντως είναι καλό νέο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ρωτάει γιατί πρέπει να αλλάξουν τα εργασιακά δικαιώματα των πολιτών που σήμερα είναι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς πρέπει να επιμείνουμε. Η στρατηγική που ακολουθούν οι κοινωτικοί εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σωστή. Δεν ξέρω αν το ίδιο από πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου. Πάντως εμείς πρέπει να επιμείνουμε για να διασφαλίσουμε μια καλή συμφωνία όσον αφορά τα δικαιώματα των πολιτών και εργασιακά και κοινωνικά. Πρέπει να υπάρξει μια καλή συμφωνία. Ένα έξυπνο και δίκαιο Brexit. Αυτά τα δύο. Έξυπνο τι σημαίνει. Σημαίνει ότι οικονομικά θα φροντίσουμε να υποφεληθούν και δύο πλευρές. Αλλά δεν θα ήταν δίκαιο αν δεν υπάρξει εγγύηση για ίσα δικαιώματα μεταξύ των μεν και των δε. Είναι λοιπόν σημαντικό να διασφαλίσουμε ένα σύστημα συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης, όπως περίπου αυτό που έχουμε σήμερα και για τους Ευρωπαίους πολίτες του σημερινούς αλλά και τους μελλοντικούς. Δεν μπορούμε να περάσουμε στο δεύτερο στάδιο των διαπραγματεύσεων αν δεν ξέρουμε ποια είναι η συμφωνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Μόνο μετά μπορούμε να μπούμε σε διαπραγμάτευση για τις μελλοντικές σχέσεις. Και μόνο έτσι μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι το Brexit θα είναι δίκαιο. Σε αυτό πρέπει να επιμείνουν οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πάνω από 5 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται σε αβεβαιότητα εξαιτία του Brexit. Και θα ήταν λάθος η στρατηγική του Ηνωμένου Βασιλείου, δηλαδή να βλέπει αυτούς οι οποίοι φεύγουν από το Ηνωμένο Βασίλειο που εκτιμάται ότι είναι ένα 20%. Και ποια είναι η ημερομηνία τώρα εξόδου. Οι Βρετανοί θέλουν από τη στιγμή που εστάλει η επιστολή για το άρθρο 50 από τον Ηνωμένο Βασίλειο, από τότε να αρχίζει να ισχύει ο χρόνος. Ενώ εγώ, και τελειώνω ο πρόεδρε, πιστεύω ότι πρέπει να μετράει ο χρόνος από τότε που γίνεται πραγματικότητα η έξοδος. Αλλιώς θα είναι σε βάρος των πολιτών. Και τέλος πάρα πολύ γρήγορα, πρέπει να διατηρηθεί η δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου και τη γνωρίζοντας το βρετανικό σύστημα μπορεί πολλοί πολίτες να μην μπορέσουν να χαίρουν των δικαιωμάτων τους. Και επίσης το θέμα της απόδειξης κατοικίας. Δεν ξέρω αν θα ζητήσουν 2, 3, 5 χρόνια πρέπει να αρχίσουν να μετράνε τα δικαιώματα αυτά. Πέρα από τα 2, 3, 5 χρόνια ότι θα τεθεί, θα πρέπει να υπάρχει ελαστικότητα και όχι λόγω γραφειοκρατίας να πλήττονται τελικά και να παραβιάζονται τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Μακιντάιρ εκ μέρου τη ομάδα CCR. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον ε, Γκίφερ Χόφστατ για αυτή την λεπτομερέστατη παρουσίαση και ενημέρωση και ε, σας ευχαριστώ για την θετική σας προσέγγιση. Πολλοί σχολιαστές ισχυρίζονται ότι στα πλαίσια του Brexit θα γίνει ένας αγώνας προς τον πάτο σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων. Εγώ δεν πιστεύω πως ε, αυτό ισχύει. Το αντίθετο μάλιστα πιστεύω πως το Ηνωμένο Βασίλειο έχει υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης, υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας από ό,τι Ευρωπαϊκή ε, Νομοθεσία. Και ελπίζω να συμφωνήσετε ότι το παρελθόν μας αποδεικνύει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζει να δεσμεύεται για την δίκαιη απασχόληση και την ασφαλή απασχόληση. Και να σας δώσω μερικά παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο στάθηκε πάνω από τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ισότητα για παράδειγμα, γονική άδεια και οι σχετικές απολαβές ίσες για όλους. Ε, ψηφίστηκε το 2014 στο Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο νόμο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κοινοτικό επίπεδο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο τα ποσοστά απασχόληση των γυναικών είναι σχετικά υψηλότερα από τον μέσο όρο τη Ένωση. 71% σε σχέση με 60% ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο στόχος είναι να φτάσουν οι γυναίκες στο 60% των ε, απολευών ε, των ανδρών μέχρι το 2020 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε πιο μπροστά από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό. Και συνεχώς λοιπόν το Ηνωμένο Βασίλειο έχει τις καλύτερες επιδόσεις ε, στην ασφάλεια στον χώρο εργασίας και από τα χαμηλότερα ποσοστά θνησιμότητα στον χώρο εργασίας επίσης. Είμαστε δεύτεροι μετά τη Μάλτα και τα ποσοστά επίσης ε, που έχουν να κάνουν με την υγεία στο χώρο εργασίας, με αναρωτικές άδειες, είναι από τα χαμηλότερα. Χαμηλά είναι επίσης τα ποσοστά ε, επισφαλούς ε, εργασίας από την πλευρά της υγείας. Το Ηνωμένο Βασίλειο λοιπόν βρίσκεται, όπως σας είπα, μπροστά ε, κανείς δεν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το Brexit ως ευκαιρία για να διαβρωθούν τα δικαιώματα των εργαζομένων και ελπίζω και εσείς να μπορέσετε να μας δώσετε τέτοιες διασφαλίσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Καλβέ Τσαμπών από την ομάδα των φιλελευθέρων. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Γκί για την παρέμβασή του. Από πλευράς των φιλελευθέρων δεν θα επαναλάβω αυτά τα οποία υπόθησαν και τα οποία με βρίσκουν σύμφωνο σχετικά με τον σφαιρικό χαρακτήρα του προβλήματος και όχι τόσο για θέματα νομοθετικά στο Ηνωμένο Βασίλειο για την προστασία των εργαζομένων. Αυτά είναι θέματα προς εμβάθυνση. Υπάρχει στήριξη λοιπόν των φιλελευθέρων στο έγγραφο του Κοινοβουλίου για το Brexit και θα το υπερασπιστούμε και στο μέλλον. Γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι στην παρούσα φάση, μετά από ένα τουλάχιστον χρόνο, δεν έχει ε, δοθεί η παραμικρή προσοχή ε, στην ε, διαδικασία αυτή. Έχουμε μπει σε μια διαδικασία εκβιασμού σε ένα θα έλεγα αιώνιο σε ένα αιώνιο καθαρτήριο το οποίο, από το οποίο δεν ξέρουμε πότε θα βγούμε. Θα ήθελα λοιπόν οι διαπραγματεύσεις ομάδες να ε, μην έχουν φόβο, να εκφράζονται ξεκάθαρα και να μην είναι υπερμετροδιπλωματικές προσωπική μου γνώμη είναι ότι δεν θα πρέπει να μην έχουμε ένα plan B ή και plan C έτσι ώστε να βάλουμε σαν στόχο μας την προστασία της ποιότητας της ζωής αν τυχόν παραταθεί ένα εκβιαστικό status quo. Η μεμονωμένες θα έλεγα αντιδράσεις δεξιά και αριστερά από τον κύριο Κάζα, από τον κύριο Γκουτιέρες ακούστηκαν. Υπάρχει μια πρόταση η οποία ξεχάστηκε λίγο και ε, εποφελούμε παρουσιάζοντάς την, είναι το θέμα των πιστώσεων των κοινοτικών ταμείων, των σχετικών με το κοινωνικό ταμείο, με το Εράσμους κτλ. Και εδώ θα πρέπει να προστατεύσουμε τη συνέχιση των προγραμμάτων αυτών και κατά συνέπεια τα δικαιώματα αυτών οι οποίοι στοχεύουν ε, σε τέτοιου είδους ε, κάλυψη ή έχουν ήδη μια τέτοια κάλυψη η οποία θα συνεχίζεται. Μια ιδέα επιπλέον. Η, θα έλεγα οι συνέπειες αυτής της πραγματικής ιστορικής ανοησίας είναι κάτι το οποίο θα θίξει ιδιαίτερα τους πολίτες της Ευρώπης και στο μέλλον. Ακόμα βέβαια δεν έχουν τελειώσει όλα. Πρέπει να εμείνουμε στα τρία κεκτημένα, δηλαδή την παρούσα συζήτηση, τη συγκυρία αν θέλετε. Είναι ε, βασικό να υπάρξουν απαντήσεις για τους πολίτες. Ε, καλό είναι να συζητήσουμε για την κατάσταση των συνόρων στο μέλλον, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει ίσως να πάρουμε και μονομερείς αποφάσεις και μέτρα για να προστατεύσουμε τους πολίτες μας. Η αξιοπιστία της δημοκρατίας στην Ευρώπη είναι υπό αμφισβήτηση. Και τελειώνοντας, η Ευρώπη θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο μας κάνει περήφανος. Ε, και σαν Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε από τη διαδικασία αυτή. Και εγώ λοιπόν προσωπικά θα ήθελα να πω ότι δεν ακτιμώ το ότι περνάμε σε κάποιες ε, διερμηνίες ε, του τι είναι ένας πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι είναι ε, το κοινωνικό όραμα κτλ. Αυτά είναι συζητήσεις οι οποίες δεν χρειάζεται να γίνουν. Νομίζω ότι θα πρέπει να ανήκει κανείς σε ένα ευρωπαϊκό κράτος μέλος δεν υπάρχουν ενδιάμεσες ρυθμίσεις και ενδιάμεσα χαρακτηριστικά καθεστώτα. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να διαπραγματευτούμε και για τους Βρετανούς, σε δύο χρόνια δεν θα διαπραγματευόμαστε για τους Βρετανούς, μια Ευρώπη πρέπει να είναι γενναιόδορη, πρέπει να είναι αλληλέγγυα και πρέπει να σέβεται τα τρία κεκτημένα σεβόμενη τα δικαιώματα των πολιτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στη Μαρτίνα Άντερσον εκ μέρους της GUNGL. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Και ακούσαμε πράγματι ότι καμία συμφωνία είναι προτιμότερη από μια κακή συμφωνία. Ακούσαμε για το κόστος ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως ε, είναι πράγματα που έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Θα ήθελα καταρχάς να ασχοληθώ με την 16η Αυγούστου που ακούσαμε ότι η Τερέσα Μέη θα προσπαθήσει να τηρήσει τη συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής, δεν θα υπάρξουν σκληρά σύνορα και όσοι μένουν στη Βόρεια Ιρλανδία όπως ε, και εγώ που έχουν δύο διαβατήρια, εγώ έχω διπλωματικό διαβατήριο και όλα θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν τα ίδια ε, δικαιώματα που απολάμβαναν μέχρι τώρα. Νομίζω πως πρέπει να τα κοιτάξουμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Νομίζω πως ε, πολλά από αυτά που ακούμε είναι ουσίας. απλά τα λένε για να τα πούν. Και πρέπει να εξετάσουμε λοιπόν ε, τις λεπτομέρειες. Νομίζω πως μας εκμεταλλεύονται και μας εκμεταλλεύονται εκβιάζοντάς μας με την Τελωνιακή Ένωση. Εάν δεν συμφωνείτε να έχουμε πρόσβαση στην Τελωνιακή Ένωση, τότε και εμείς θα καταστρέψουμε τη συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. Θα υπάρξει σκληρό σύνορο ε, στην Ιρλανδία κτλ. κτλ. Και νομίζω πως ε, πολλοί ε, δεν έχουν ακριβή εικόνα του τι συμβαίνει. Νομίζω πως είμαστε απερίσκεπτοι, πως παίζουμε με τη φωτιά. Είναι η Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής, μια συμφωνία που ε, αποκτήσαμε μετά από πολλούς αγώνες, με αίμα σχεδόν και πρέπει να την προστατεύσουμε. Ας μην ξεχνάμε τα δικαιώματα των πολιτών. Ας μην ξεχνάμε το ένα εκατομμύριο ε, πολιτών που ζει στη Βόρεια Ιρλανδία, που έχει την πολυτέλεια, πολυτέλεια θα πω αυτή τη στιγμή, να έχει Ιρλανδικό διαβατήριο. Ε, όταν κάποιοι άλλοι, ε, όταν κάποιος ζει στην Γερμανία, ε, θεωρείται Ευρωπαίος πολίτης, αλλά τα πράγματα αλλάζουν για την Ιρλανδία. Αν πάρουμε δηλαδή τις μετρητής αυτά που είπαν για τους Ιρλανδούς πολίτες, μιλάμε για το άρθρο 9, για την ίση μεταχείριση όλων των πολιτών, άρθρο 10, δικαίωμα ψήφου. Αλλά θα ολοκληρώσω λέγοντα ε, τα εξή, γιατί ξέρω πώ υπάρχουν και άλλοι που θέλουν να μιλήσουν, ότι στα πλαίσια τη συμφωνία τη μεγάλη παρασκευή, ε, όπως αυτή είναι ένα διεθνέ έγγραφο που έχει συζητηθεί και στα πλαίσια των ΗΠΑ πρέπει να διασφαλιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα τηρήσει τι υποχρεώσει του άρθρου 5, που ε, αναφέρει ότι δεν πρέπει να θέσει σε κίνδυνο οποιαδήποτε διεθνή συμφωνία και να μην... Ε, κινδυνεύσει η ειρηνευτική διαδικασία, να μην κινδυνεύσουν όλα αυτά που έχουμε επιτύχει μέχρι τώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θεωρώ πως πρέπει να ε, ζητήσει από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου κάποια διασφαλίσει διότι μπορεί να έχουν πει μεν πολλά, αλλά θεωρώ πω δεν έχουν κάνει τίποτα άλλο από το να εκμεταλλευτούν τι περιστάσει. Και η κυβέρνηση τη Ιρλανδία έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν πρόκειται να δουλέψει ε, προ το συμφέρον εκείνων που θέλουν το Brexit. Ελπίζω να τηρήσει αυτέ τι υποσχέσει που έδωσε και να κρατήσει το λόγο τη. Θα ήθελα λοιπόν να σα ευχαριστήσω κλείνοντα για την παρουσίαση και να πω ότι ελπίζω το Κοινοβούλιο να παραμείνει ε, πίσω από την δήλωσή του, πως θέλει δηλαδή να στηρίξει τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής ε, με όλες τις, τις λεπτομέρειες. Ευχαριστώ πολύ. κύριε κυρία Ράιντ και εκ μέρους των Πρασίνων έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου για αυτήν την λεπτομερή παρουσίαση. Να πω πως συνεχίζω να θεωρώ ότι είναι λάθος όλα αυτά που συμβαίνουν και θα το πω ευθέως, ε, παρά τα όσα μας είπατε, νομίζω πως και κυριαρχεί ένα χάος και αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να συμμαζέψουμε τα σημάζευτα, αν θέλετε. Υπάρχουν πολλά διευκρίνηστα σημεία Ήλπιζα να ακούσουμε περισσότερα λεπτομέρειε επί του περιεχομένου, να ακούσουμε περισσότερα για τη δομή και αυτόν θέλουμε να πάμε μπροστά, να προχωρήσουμε, γιατί πολύ μου άρεσαν αυτά που άκουσα για το ότι χρειαζόμαστε μια νέα συμφωνία, ότι οποιαδήποτε συμφωνία είναι καλύτερη από το να μην υπάρχει καθόλου συμφωνία, αλλά εάν υπάρχει ακόμα αυτό το μπέρδεμα, γίνεται κάτι, γίνονται προετοιμασίες και τι θα γίνει σε περίπτωση που δεν καταλήξουμε σε συμφωνία. Αυτό λοιπόν το μπέρδεμα είναι ένας λόγος ε, για να παραμείνω στο Κοινοβούλιο όταν θα ξαναζητήσει το Ηνωμένο Βασίλειο να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έρθει αυτή η ώρα. Έχω όμως κάποιες ερωτήσεις. Μας είπατε ότι λαμβάνετε πολλές επιστολές από Βρετανούς πολίτες αλλά και από πολίτες της Ένωσης που αναφέρουν τις ανησυχίες τους για το τι θα γίνει, τι θα περιέχει αυτή η συμφωνία. Εγώ θέλω να, ρωτήσω, ε, να ζητήσω μάλλον οι ανησυχίες των Ευρωπαίων πολιτών να μην χρησιμοποιηθούν ως διαπραγματευτικό χαρτί. Υπάρχουν πολλοί πολίτες οι οποίοι ζουν σε άλλη χώρα, έχουν κάνει την άλλη χώρα νέα τους πατρίδα και τώρα πρέπει να ε, βρουν έναν τρόπο να ξεφύγουν από αυτό το μπέρδεμα. Τώρα έχω μία ερώτηση σχετικά με τους αυτοαπασχολούμενους και τους επιχειρηματίες. Έχει δοθεί προτεραιότητα σε αυτές τις ομάδες και αυτό είναι κάτι το οποίο οραματίζεστε να επαναλάβετε και στα πλαίσια της συμφωνίας του Brexit. Μετά, αποσπασμένοι εργαζόμενοι. Αυτή τη στιγμή συζητούμε την ανανέωση της οδηγίας για την απόσπαση εργαζομένων. Βασίζεται στην ελευθερία της παροχής υπηρεσιών, αλλά αφορά μέσα και τα δικαιώματα των πολιτών. Γι' αυτό λοιπόν η ερώτησή μου ε, έχει να κάνει με το τι θα γίνει από εκεί και στο εξή. Και τέλος, πολύ συχνά ακούμε πως όλες οι κυβερνήσεις και των 27 κρατών μελών είναι ενωμένε, είναι με μία φωνή. Θα ήθελα λοιπόν κάποια παρασκηνιακά σχόλια. Αυτό ε, ισχύει, αληθεύει, τι γίνεται, τι ακούτε στα, παρασκηνία, ποιος είναι ο, ρόλος του Κοινοβουλίου και πώς μπορεί να διατηρήσει αυτήν την ενότητα. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ρέιμοντ Φίντς έχει το λόγο εκ μέρους του EFTD. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα κύριε Φερχόφστατ. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ένα τεράστιο εμπορικό έλλειμμα απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χρειάζεται την αγορά της ε, την αγορά της. Πολλές θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτώνται από το Ηνωμένο Βασίλειο και ε, το Ηνωμένο Βασίλειο μάλιστα έχει μια οικονομία που είναι τόσο δυνατή όσο οι, πιο, οι 20 πιο αδύναμες ε, οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς λοιπόν μπορούμε να εξηγήσουμε στους Ευρωπαίους πολίτες ότι χάσαν τις δουλειές τους γιατί απέτυχε το ε, κίνημα του φεντεραλισμού. Πώς μπορούμε να τους εξηγήσουμε ότι θέλουν μια Ευρώπη πάση θυσία και θα θυσιάσουν και την οικονομική σταθερότητα η συμφωνία με, την, ε, με το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι προς το συμφέρον των Ευρωπαίων εργαζομένων. Πρέπει να είναι προς το συμφέρον όλων των πολιτών και όχι μόνο προς το συμφέρον της, ε, του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Κάποιο συνάδελφος είπε νωρίτερα πως ε, το Κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου ήδη έχει ανώτερη νομοθεσία για εργασιακά θέματα και θα συνεχίσει να έχει όταν αποχωρήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σύμφωνα με την Bruegel που είναι μια think tank ε, υπέρ της Ευρώπης υπάρχει ένα ε, ποσό 133 δισεκατομμυρίων το οποίο ε, θα κληθεί το Ηνωμένο Βασίλειο να επιστρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως κομμάτι του, των όρων του διαζυγίου. Οποιαδήποτε συμφωνία όμως ε, που περιλαμβάνει ρήτρε τέτοιου είδους, ε, να είστε σίγουροι πως θα καταψηφιστεί από το Βρετανικό Κοινοβούλιο και έτσι θα είμαστε ελεύθεροι, ευτυχισμένοι και ανεξάρτητοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, Ντομινίκ Μαρτάν τώρα από το ΙΕΝΕΦ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο κύριε Μαρτάν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ τον συντονιστή. Φοβάμαι. Και φοβάμαι γιατί ακούω από εδώ και από εκεί σκληρά λόγια. Είναι καταστροφή για τον Αμένο Βασίλειο, λένε. Μετά τα είχαμε από δημοσκοπήσεις και αναλύσεις. Είναι σφάλμα. Αν ξαναψήφιζαν, θα ξαναψήφιζαν αλλιώς. Ε, δεν διαβάζουμε τις ίδιε δημοσκοπήσει, δεν έχουμε τις ίδιε αναλύσεις. Όσον αφορά την απασχόληση και τα κοινωνικά ζητήματα συγκεκριμένα, θα θέλανε, θα θέλατε, πολύ εδώ τέλο πάντων θα ήθελαν να κάνουμε σαν να μην συνέβη τίποτα απολύτως. Σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα απολύτως. Και πρέπει οπωσδήποτε να διατηρήσουμε την ίση μεταχείριση. λες και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπήρχε ζωή. Λες και εκτός αυτής της Ένωσης δεν υπάρχει μέλλον. Μα αγαπητοί συνάδελφοι, να σας θυμίσω ότι στον πλανήτη αυτό που ζούμε υπάρχουν χώρες, δεκάδες χώρες, πολύ περισσότερες από τις 27 δηλαδή, που ζουν και έχουν μια αυτοκρατορία εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός Σέγγεν ή και μέσα στο Σέγγεν. Ελβετία, μια πολύ μικρή χώρα, η οποία τα καταφέρνει μια χαρά. Και έτσι, είπατε 29 Σεπτεμβρίου 2009, πριν το δεύτερο γύρο της ψηφοφορίας στην Ιρλανδία, είπατε ότι η Λισαβόνα θα έχει δικαιώματα βάση του άρθρου 50. Αυτή θα είναι η νομική βάση. Έτσι είχατε πει. Τώρα ξέρω ότι σας περιπλέκει τη ζωή. Με ισχυρή νομική βάση για να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των εργαζομένων, όπως εκείνο στις ε, συλλογικέ συμβάσεις και άλλα, και ότι δεν μπορεί να υπάρχει dumping εφόσον επικυρωθεί η συνθήκη της Λισαβόνας. Αυτά λέγατε. 29 Σεπτεμβρίου Τώρα το κοινωνικό dumping είναι η οδηγία για τους αποσπασμένους. Μα κύριε Σιτονιστέ τότε πώς τα είχατε προβλέψει όλα αυτά. Τώρα, μετά τη δεύτερη ψηφοφορία στην Ιρλανδία, τι είπατε, κατά λέξη, είπατε. Σήμερα είναι μια υπέροχη μέρα για την Ευρώπη αυτή. Σήμερα είναι η πρώτη μέρη ενός ε, νέου μέλους για μια δημοκρατική Ευρώπη με αυτή τη νέα συνθήκη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορεί να αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα όπως οικονομική και δημοσιονομική κρίση με αποτελεσματικό και συντονισμένο τρόπο. Το 2009 αυτά, έτσι, λίγο μετά το 2008. Τώρα είμαστε σχεδόν 10 χρόνια αργότερα και πάλι τα είχατε προβλέψει και λέγατε ότι η Ευρώπη θα μιλούσε με μία φωνή στον κόσμο και θα έδινε τις απαντήσεις που αναμένουν από αυτήν οι πολίτες. Αυτά είπατε τότε. Συγγνώμη που σας βάζω μπροστά στα δικά σας τα λεγόμενα, αλλά έχει σημασία. Και τέλος, μια που η δημοκρατία είναι μια λέξη που έχετε συνέχεια στο στόμα, να ξέρετε ότι πριν από λίγο πάνω από ένα χρόνο, εκατομμύρια 17.142.000 και κάτι Βρετανοί ψηφοφόροι είπαν όχι. Εδώ ή οπουδήποτε αλλού κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων μπορείτε σας παρακαλώ να το έχετε υπόψη σας ότι υπάρχει ελευθερία των λαών στην αυτοδιάθεση. Κύριε συντονιστά. Σα ζητάω λοιπόν περισσότερη μετριοπάθεια και περισσότερη ταπεινοφροσύνη. Ευχαριστώ κύριε συντονιστά. Σας ευχαριστώ. Έχω άλλους επτά εγγεγραμμένους που θέλουν να θέσουν ερωτήματα προς τον κύριο Φερχώστατ. Θα επανέλθουμε στους υπόλοιπους γιατί καιρός είναι ο κύριος Φερχώστατ να ξεκινήσει να αντιδρά και να διευκρινίζει ε, τα θέματα που έθεσαν αυτοί που κατέθεσαν τις ερωτήσεις τους. Ευχαριστώ Πρόεδρε για την τελευταία παρατήρηση για τα 17 εκατομμύρια. Αν κατάλαβα καλά υπάρχουν άλλα 45 εκατομμύρια που είπαν ναι ή που δεν εκφράστηκαν. Έχω σπουδάσει νομική, αλλά τα μαθηματικά δεν είναι και πάρα πολύ δύσκολα. Αν 17 εκατομμύρια είπαν ότι πρέπει να φύγουν, 45 ε, εκατομμύρια δεν είπαν τίποτα και κάποιοι είπαν να μείνουν. Μπορούμε να τα συζητήσουμε τα θέματα αυτά όσο θέλετε. Αλλά εγώ σέβομαι την απόφαση του Βρετανικού λαού, πρέπει να γίνει σεβαστή και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να δώσουμε περιεχόμενο και νόημα στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας που προηγήθηκε και αυτό προσπαθούμε ακριβώς να πετύχουμε με τις διαπραγματεύσεις για τον κύριο Φίντσα. Ε, Είπατε ότι εμείς τους πετάξαμε έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, δεν είναι ακριβώς έτσι. Μόνοι τους αποφάσισαν να φύγουν. είναι μια κυρίαρχη δική τους απόφαση. Γιατί λέτε ότι εσείς δεν κάνατε αυτό, δεν κάνατε το άλλο, δεν λάβατε υπόψη σας το ένα, δεν λάβατε υπόψη σας το άλλο. Δεν λάβατε υπόψη σας το ότι μπορεί να χάσει η υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση ή τους διώξατε. Ε, όχι, δεν τους διώξαμε, μόνοι τους αποφάσισαν να φύγουν. Αν είναι σωστή η απόφαση αυτή, αυτό δεν θα το πω εγώ. Εγώ βλέπω πώς πηγαίνει η στερλίνα, εγώ βλέπω τι γίνεται με τον πληθωρισμό. Βλέπω επίσης και ότι ορισμένες, ορισμένα πολιτικά κόμματα σκέφτονται τώρα ποιες είναι οι οικονομικές συνέπειες μιας τέτοιας απόφασης. Πάντως, είναι σαφές ότι τις ευθύνες μας σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να τις αναλάβουμε. Έρχομαι τώρα στις δύο πρώτες παρεμβάσεις από τους συντονιστές του ΕΛΚ και των σοσιαλιστών. Το βασικό πρόβλημα με την πρόταση για τα δικαιώματα των ε, πολιτών από όλες τις πλευρές δεν είναι μόνο το ότι το καθεστώς αυτό του τακτοποιημένου πολίτη μειώνει τον αριθμό των δικαιωμάτων που προτείνει το Ηνωμένο Βασίλειο. περίπου καλύπτει τα ισχύοντα δικαιώματα με μια μεγάλη ίσως εξαίρεση, δηλαδή την οικογενειακή επανένωση, όπου εκεί υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση ανάμεσα στο τάτους κβο, στη σημερινή κατάσταση και ποια θα είναι τα δικαιώματα αυτά μετά από την εισαγωγή του καθεστώτος του τακτοποιημένου πολίτη. Το βασικό πρόβλημα είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να πάρει κανείς το καθεστώς αυτό. Πρέπει να καταθέσει μία αίτηση, θα ακολουθήσει μία διαδικασία, ε, αξιολόγησης, ε, πληρωμή, διοικητικά και γραφειοκρατικά άχθη. Θα πρέπει να το κάνουμε ξεχωριστά για κάθε μέλος της οικογένειας, ε, δεν μπορούμε να το κάνουμε για την οικογένειά μας, πρέπει ο καθένας να κάνει για τον εαυτό του κτλ. Το βασικό πρόβλημα λοιπόν είναι το περιεχόμενο, περιορίζονται τα ισχύοντα δικαιώματα, τα υπόλοιπα περίπου καλύπτονται. Και το θέμα είναι η διαδικασία που δημιουργείται. Εμείς αντίθετα λέμε ότι ξέρουμε ποιοι είναι οι πολίτες της Ένωσης που ζουν στη Μεγάλη Βρετανία και θα πρέπει ακριβώς να εγγυηθούμε τα δικαιώματά τους. Και όχι ξαφνικά να πούμε «Α, ναι, υπάρχουν 3 εκατομμύρια που ζουν εκεί και από εδώ και πέρα θα πρέπει να κάνουν αιτήσει ο καθένας ξεχωριστά και να αποδείξουν το εξή ο καθένας με διαφορετικό τρόπο». Έχουμε να κάνουμε με μια μεγάλη λοιπόν διαφορά απόψεων αυτό. Είναι αλήθεια ότι η πρόταση των Βρετανών καλύπτει το 85% των δικαιωμάτων. Αλλά δεν είναι αυτόματο, πρέπει να το ζητήσει κανείς για να το αποκτήσει, Εδώ σήμερα το έχουν το καθεστώς αυτό. Εν πάση περιπτώσει προσπαθώ να εξηγήσω ποιες είναι οι βασικές δυσκολίες που καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε. η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου θα πρέπει να γίνεται σεβαστή και όπως είπα δεν θα θέλαμε ο καθένας από εδώ και πέρα ε, σε ένα ατομικό φάκελο να κάνει αιτήσει, να λέει ακριβώς ε, τι χρειάζεται να γίνει από εδώ και πέρα και ποιες είναι οι διαδικασίες μέσα από τις οποίες πρέπει να περάσει, που δεν υπάρχουν σήμερα. Για την κυρία Μάκεντάιρ και κάποιος άλλος αναφέρθηκε επίσης για ένα plan B. Εγώ ξεκίνησα από την ιδέα ότι αυτό το οποίο απαιτείται είναι οι διαπραγματεύσεις και πρέπει να υπάρξει μια λύση. Είναι σαφές ότι αν κάτι τέτοιο δεν συμβεί και αν ε, δεν ε, ε, δώσουν λύσεις οι διαπραγματεύσεις αυτές θα πρέπει να βρούμε άλλη λύση. Αλλά ξεκινώ με την προϋπόθεση ότι οι διαπραγματεύσεις προχωρούν και είμαστε σε θέση να καταλήξουμε σε μια συμφωνία επί της ουσίας για τη νέα αυτή σχέση. Αλλά δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε τα θέματα αυτά αν δεν υπάρξει σημαντική πρόοδος στα πλαίσια της Συμφωνίας Εξόδου. Για η Συμφωνία Εξόδου προβλέπεται στις συνθήκες. Και στις συνθήκες λέμε ότι θα πρέπει να γίνει Συμφωνία Εξόδου σε σχέση με τον καθορισμό της νέας σχέσης. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια βασική, θέλετε, αντίληψη ε, για μια καθορισμένη νέα εταιρική σχέση. Και όπως ξέρετε κυρία Μάκεντάιρ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ξεκαθαρίσει εδώ, ίσως είναι το μόνο θεσμικό όργανο, που λέει ότι θα πρέπει ίσως μέσω μιας συμφωνίας σύνδεσης να δούμε τους τρόπους συνεργασίας με το Ηνωμένο Βασίλειο. Γιατί μια τέτοια συμφωνία δεν είναι μόνο μια συμφωνία για το εμπόριο και την οικονομία, αλλά και για άλλα θέματα, όπως η συνεργασία στην έρευνα, στον πολιτισμό, στην άμυνα στις εξωτερικές υποθέσεις κτλ. Τώρα για την κυρία Άντερσον και τη Βόρεια Ιρλανδία. Νομίζω εδώ ότι είναι εύκολο να μιλάει κανείς για τη Βόρεια Ιρλανδία, είναι δύσκολο να βρει λύσεις όμως. Εμείς δεν θέλουμε σκληρά, κλειστά ή ημίσκληρά ε, και κλειστά σύνορα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το διευκρινίσουμε. Αυτή τη στιγμή δεν αποκλείουμε τίποτα. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε και που είπαμε τις τελευταίες εβδομάδες είναι ότι δεν πρέπει να δώσουμε την απόφαση ε, ότι υπάρχει μια αόρατη ομάδα, υπάρχουν αόρατα σύνορα. Αν είναι αόρατα δεν είναι σύνορα. Εγώ έχουμε από την περιοχή του Μαγκρίτ, ξέρετε τον πίνακα του Μαγκρίτ που λέει ότι αυτό δεν είναι μία πίπα. Έτσι λέει ο πίνακας. Είναι λίγο σουρεαλιστικό αυτό. Ε, λένε οι Βρετανοί λοιπόν ότι κοιτάξτε έχουμε σύνορα που δεν είναι σύνορα. Ε, δεν γίνεται. Αν δεν φαίνονται τότε δεν είναι σύνορα. Και στην ευρωπαϊκή ιστορία θα έλεγα ε, δεν υπήρχαν μερικές φορές σύνορα. Το 18ο αιώνα ήταν εύκολο να φτάσει κανείς από το... όταν πήγε ο Μοντένιε στην Ιταλία, δεν τον σταμάτησαν στα σύνορα και δεν ε, είχε διαβατήριο να δείξει. Συνεπώς λοιπόν υπήρχε κάποτε Ευρωπαϊκή Ήπειρος χωρίς σύνορα, δεν έχουμε να κάνουμε με κάτι καινούριο. Τα σύνορα προήλθαν από τον 19ο αιώνα, είναι εφεύρεση του 19ου αιώνα και καλό θα είναι να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε ότι τότε αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε αυτή τη γραφειοκρατική αν θέλετε διαδικασία. Εν πάση δεν ξέρω γιατί τα λέω αυτά, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα σύνορα είναι σύνορα όταν υπάρχουν και τα σύνορα όταν δεν υπάρχουν δεν είναι σύνορα. Είναι ένας πίνακας του Μαγκρίτ που ζωγραφίζει μια μικρή πίπα και λέει αυτό δεν είναι μια πίπα. Συνεπώς λοιπόν δεν είμαι 100% σίγουρος και το λέω αυτό με κάθε ειλικρίνεια ότι είναι σωστές οι προτάσεις της Βρετανικής κυβέρνησης. Όχι, δεν μπορώ να τις δεχτώ. Νομίζω ότι απαιτείται περισσότερη φαντασία για να βρούμε μια κάποια λύση. Και βλέπετε ότι είμαι πολύ προσεκτικός όταν το λέω αυτό. Για την κυρία Ράινκια και το λεγόμενο ring fencing. Κοιτάξτε, η συμφωνία αποχώρησης έχει τρία τμήματα. Το μεθοριακό θέμα, την οικονομική ρύθμιση ε, και τα δικαιώματα των πολιτών. Θέση του Κοινοβουλίου είναι ότι θέλουμε να υπάρξει πρόοδος στα δικαιώματα των πολιτών. Και όταν καταλήξουμε σε μια συμφωνία εκεί, τότε θα είναι τμήμα της συνολικής συμφωνίας. εμείς θα πρέπει να εγκρίνουμε τη συμφωνία αυτή. Αν είναι μια συμφωνία απλή αποχώρησης, φυσικά εμείς θα πούμε όχι. Και τότε μόνο από εκεί και πέρα θα ισχύσει. Αλλά συμφωνώ μαζί σας ότι όχι ρήτρε προστασίας, ring fencing δηλαδή. Αν έχουμε μια συμφωνία και μπορούμε να δώσουμε νομική βεβαιότητα στους πολίτες, ας το κάνουμε από τώρα. Και εμείς περιμένουμε το 19 να δούμε τι θα κάνουμε. Ας μην περιμένουμε το Μάρτιο του 2019 για να βρούμε μία πρόταση. Δεν είναι κάτι το σωστό αυτό. Εάν υπάρχει επαρκής πρόοδος λοιπόν και αν τους επόμενους μήνες η πρόοδος αυτή χαρακτηριστεί και από πρόοδο στα δικαιώματα των πολιτών, έχουμε την υποχρέωση να το παρουσιάσουμε αυτό στους Ευρωπαίους πολίτες και να μην περιμένουμε το Μάρτιο του 2019 πριν υιοθετήσουμε επίσημα τη συγκεκριμένη πρόταση. Αυτά. Και το έχω πει επανειλημμένα σε όλους όσους και σε όλες τις πολιτικές ομάδες και κινήσεις που δημιουργήθηκαν και στο Ηνωμένο Βασίλειο και εδώ, ότι αυτός είναι ο βασικός μας στόχος, το ταχύτερο δυνατόν ασφάλεια για τους Ευρωπαίους πολίτες. Και όλα αυτά θα πρέπει να πάρουν το πράσινο φως από το Κοινοβούλιο το 19. Και πρέπει να υπάρχει και ενότητα ανάμεσα στους 27. Δεν είναι δική μου δουλειά να το κάνω αυτό. Αλλά είναι αλήθεια ότι το Κοινοβούλιο παίζει εδώ κάποιο ρόλο. Νομίζω ότι έχουμε ίσως κάποιες ιδεολογικές διαφορές σε επίπεδο Ευρώπης. Ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο αντιπροσωπεύει απλά τα εθνικά του συμφέροντα. Ανεξαρτήτως λοιπόν του τι λέμε για τον Brexit, το κάτι το θετικό είναι ότι έχει δημιουργήσει θα έλεγα ε, μια τάση αν θέλετε ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή Ενότητα, την Ευρωπαϊκή Ιδέα. Ε, βλέπουμε πραγματικά να αυξάνεται η εμπιστοσύνη των λαών στην ευρωπαϊκή προσπάθεια. Η εντύπωσή μου είναι λοιπόν ότι έχει δημιουργήσει αν θέλετε το Brexit μεγαλύτερη ενότητα από τις προσπάθειες επικοινωνίας που κάναμε στο παρελθόν. Λοιπόν, ίσως να είναι υπερβολική αισιοδοξία μου. Δεν έχω να πω κάτι άλλο σε αυτή τη φάση. Υπέροχα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι μπορούμε να συνεχίσουμε με τις υπόλοιπες ε, ερωτήσεις, τους υπόλοιπους ε, συναδέλφους στον κατάλογο. Και θα δώσω το λόγο στον κύριο Τόμας Μάν. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραίο όνομα έχετε. Χαίρομαι πάρα πολύ λοιπόν κύριε Φερχόφστατ που εσείς έχετε αναλάβει την ευθύνη γιατί είστε ένας από αυτούς που έχουν όρεξη για κουβέντα. Δεν ε, μας λέτε βαρετά πράγματα, μιλάτε έντιμα μέσα από την καρδιά σας. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ που είστε εσείς και που ήρθατε ε, σήμερα. Αυτό θέλουμε, ανθρώπους σαν και εσάς που θέλουν αποτέλεσμα. Αυτό πρώτον. Δεύτερον, ε, χαίρομαι πάρα πολύ που η Τερέζα Μέη απέτυχε παταγωδώς ε, να περάσει αυτά που θέλει. Να περάσει αυτά που θέλει ακριβώς γιατί υπήρχαν αυτοί οι νέοι που ε, αντιστάθηκαν. Και ελπίζω οι νέοι και στη δική μου χώρα να συμμετέχουν στις εκλογές. Τώρα, κοινωνική προστασία. Εδώ με βρίσκεται απόλυτα σύμφωνο. Πολλές φορές έχω λάβει πληροφορίες από πολίτες οι οποίοι μου λένε ότι από τότε που ελήφθη αυτή η λάθος για μένα απόφαση μας εκμεταλλεύονται. Μας εκμεταλλεύονται στο έπακρο. Και τώρα λένε πως δεν θέλουν τους ε, ξένους, δεν θέλουν τους ξένους εργαζόμενους, όμως ε, ε, η αλήθεια είναι ότι αυτές οι ομάδες που είναι κυρίω Πολωνοί, κάθε άλλο παρά ανεπιθύμητοι ήταν. Τους ήθελαν, του έφεραν, τους κάλεσαν. Γι' αυτό λοιπόν η κοινωνική ασφάλεια και αυτές οι, ε, αυτά τα επιχειρήματα είναι λόγια του αέρα. Τώρα, πρέπει να συζητήσουμε κάποια πολύ σημαντικά θέματα. Διαμεθοριακούς εργαζόμενου. Υπάρχει η σχετική οδηγία την οποία πρέπει να ακολουθήσουμε, πιστεύω. Τώρα, τι γίνεται με του διαμεθοριακούς εργαζόμενου από τη Βόρεια Ιρλανδία στην Ιρλανδία. Σίγουρα πρέπει να προστατευτεί η ειρήνη στην περιοχή, η ειρηνευτική διαδικασία και να, ε, να φροντίσουμε να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα αυτών των εργαζομένων. Γνωρίζουμε περί τίνος πρόκειται. Όμω, ε, τι γίνεται στην περίπτωση που μια χώρα δεν είναι πλέον μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, εδώ αλλάζουν τα πράγματα, θα αλλάξουν τα σύνορα. Πώς μπορούν ε, να γίνονται έλεγχοι στα σύνορα. Να τονίσω εδώ πως υπάρχει θέμα, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να τεθεί σε κίνδυνο η ειρηνευτική διαδικασία, να ξαναυπάρχει πόλεμο στην περιοχή. Θεωρώ πως είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Φερχόφστατ, το πρώτο ε, σχόλιο σας, δηλαδή ε, να υπάρχει πλήρη επίγνωση για το ποιο είναι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι βουλευτές πρέπει να συμμετέχουν. Θέλουμε διαφάνεια. Μας μιλήσατε για το χρονοδιάγραμμα, μας μιλήσατε και για σύγχυση. Αυτή η σύγχυση όμως οφείλεται στο ότι δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Δεν ξέρουμε τι γίνεται εδώ, δεν ξέρουμε τι θα κάνει η κυρία Μέη, δεν ξέρουμε αν θα παραμείνει ο κύριο Ντέιβι υπεύθυνο ε, ε, Brexit. Όμως, δεν ξέρουμε τι γίνεται από την πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου, ξέρουμε όμω ότι εδώ έχουμε τον ε, κύριο Μπαρνιέ, ο οποίο είναι ένα σταθερό άνθρωπο τον οποίο μπορούμε να στηριχτούμε και αυτή η σταθερότητα από τη δική μα πλευρά σίγουρα θα βοηθήσει σημαντικά. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Μαν. Θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους να περιορίσουν το χρόνο του ομιλίας τους στα δύο λεπτά. Το λόγο έχει ο επόμενος συνάδελφος. Σας ευχαριστώ πολύ λέει ο κύριος Σάιμον. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φερχόφστατ που ήρθατε. Εγώ εκπροσωπώ την περιοχή των Δυτικών Μίτλαντς, 6,5 εκατομμύρια πολίτες δηλαδή, στην κεντρική Αγγλία και το συμφέρον των ε, πολιτών νομίζω πως ε, δεν αναγνωρίζετε και δεν εκπροσωπείτε από την Βρετανική κυβέρνηση. Εμείς είμαστε μια μεταποιητική, μια περιοχή που ασχολείται με τη μεταποίηση, με την ανώτατη εκπαίδευση, με τομεί οι οποίοι δεν είναι καθώς φαίνεται σημαντικοί για το Ηνωμένο Βασίλειο, για την κυβέρνηση της ε, Τερέζα Μέη. Εξάγουμε πολλά προϊόντα στην Κίνα και η περιοχή των Δυτικών Midlands είναι μια από τις ε, περιοχές με τη μεγαλύτερη πολυμορφία στον κόσμο. Αυτό βέβαια είναι κάτι που αγνοεί παντελώς η κυβέρνηση των συντηρητικών εκεί. Είμαστε λοιπόν μία από τις ε, ελάχιστες ε, περιπτώσεις που έχουμε διαφορετική στάση. Και θα ήθελα λοιπόν εδώ να ρωτήσω εσάς, εάν υπάρχει κάποιος χαρακτηρισμός που μπορείτε να δώσετε στην προσέγγιση της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου για τις διαπραγματεύσεις που να ε, αντικατοπτρίζει την πολυμορφία που χαρακτηρίζει τη χώρα μου. Κάποια περιφερειακή διάσταση, οτιδήποτε που να δείχνει την ε, διάσταση της ε, ολόκληρης της χώρας και που δεν είναι ε, κυριευμένο από το Λονδίνο. Κάτι που φαίνεται και δείχνει όλη την επικράτεια της χώρας μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βασίρη έχει το λόγο. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Φερχόστατ για την παρουσίασή του. Αλλά όταν μιλάμε για φόβους για μετά το Brexit των εργαζομένων, είναι κάτι που κάτι που στρεβλώνει. Το Brexit δεν πρέπει να είναι ευκαιρία για μείωση δικαιωμάτων, μείωση της προστασίας των ε, ξένων εργαζομένων στις χώρες μας. Σε αυτά τα πράγματα εμείς είμαστε πιο μπροστά και πιστεύω ότι θα παραμείνουμε έτσι. Το Ηνωμένο Βασίλειο ηγείται στην Ευρώπη όσον αφορά τις προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Μάλλον ε, Άλλοι έχουν να μάθουν από εμά για την ίση μεταχείριση των γυναικών και για την ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Αν νομίζετε ότι ο κόσμος θα γυρνάει μόνο αν η Ευρωπαϊκή Γραφειοκρατία το πει, εσφάλετε, γιατί θα συνεχίσουμε να ζούμε και χωρίς αυτούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε όταν ήσασταν σύντομος. Η κυρία Ρανσαρτιέ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ και σας Πρόεδρε για την παρέμβασή σας. Μας διευκρινίσατε ποιες είναι οι μέθοδοι εργασίας σας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ επίσης που φροντίζετε να υπάρχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτήν την διαπραγμάτευση για τον Brexit. Μερικές φορές το ξεχνάμε ότι είναι σημαντικό. Μία ερώτηση έχω. Και εμεί εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δουλεύουμε πάνω στην οδηγία για τους αποσπασμένους εργαζόμενους και ελπίζουμε και εμεί να καταλήξουμε σε μια εξέλιξη τη οδηγίας αυτή, να υπάρξει αναθεώρησή τη. Πολύ εδώ ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Μπορείτε λοιπόν να μας πείτε εσείς πώς θα λάβετε υπόψη σας μια τέτοια εξέλιξη, γιατί ο συνάδελφος Τόμας Μαν αναφέρθηκε στους Πολωνούς, εντάξει, Υπάρχουν οι Πολωνοί στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά υπάρχουν και Βρετανοί σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες σε μεγάλους αριθμούς και τους χρειαζόμαστε και αυτούς. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Μωρό Σατιέ. Γιάννα τον, παρακαλώ Γιάννα. Ευχαριστώ Γκί για την παρουσίαση αυτή. Δύο πράγματα θέλω να διευκρινίσω. Μιλάμε για τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών αλλά έχουμε και Ευρωπαίους μη πολίτες. Στην Εστονία και στην Λετωνία, για παράδειγμα, υπάρχουν πολλοί που θα έχουν πρόβλημα, που και τώρα έχουν πρόβλημα, και αν δεν τους λάβουμε υπόψη μας, στο μέλλον θα έχουν ακόμα μεγαλύτερα. Και κάτι άλλο για την εργασία. Είπατε ότι υπάρχει μια ομάδα εργασίας και μια διευθυντική ομάδα. Ξέρετε όμως ότι υπάρχουν και επιτροπές ελέγχου που έχουν ε, φτιαχτεί ε, στο πολιτισμό για παράδειγμα. Οπότε εμεί δεν καταλαβαίνουμε πολύ καλά πώς πρέπει να προχωρήσουμε με αυτές τις δομές. Υπάρχουν οι ομάδες ελέγχου και υπάρχουν και άλλες που μας αναφέρατε εσείς. Πώς θα συνεργαστούν όλοι αυτοί μεταξύ τους. Η κυρία Γιουγκέριος τώρα. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ για την παρουσίαση. Και μετά από όλες αυτές τις ερωτήσεις, εμένα μου μένουν δύο ζητήματα. Υπάρχουν πολλοί Βρετανοί που λένε τα εργασιακά δικαιώματα στον Ηνωμένο Βασίλειο είναι καλύτερα από ό,τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε μήπως εμείς να πάμε να ενταχθούμε στην, ε, στον Ηνωμένο Βασίλειο για να έχουμε καλύτερα εργασιακά δικαιώματα. Παρόλο που εγώ ξέρω ότι τα τελευταία χρόνια όλη η κοινωνική πρόοδος έχει εμποδιστεί από τους Βρετανούς ευρωβουλευτές. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι, το είπε και η κυρία Μαρανσατιέ για την οδηγία για τους αποσπασμένους και ο συντονισμός της κοινωνικής ασφάλισης με απασχολεί στη νέα πρόταση. Τον Οκτώβριο θα έχουμε ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα δικαιώματα των πολιτών. Τι θα γίνει με αυτές τις δύο υποθέσεις που και εσείς είπατε ότι είναι σημαντικές για τα δικαιώματα των πολιτών. Και τον Οκτώβριο, όσο θα προχωράμε στην εξέλιξη αυτών των δύο υποθέσεων, τι θα γίνει ο κύριος Φεχάστατ να απαντήσω αμέσω στις τρεις αυτές ερωτήσεις που αφορούν το ίδιο θέμα για την απόσπαση των εργαζομένων. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν αποτελεί μέρος της συμφωνίας αποχώρησης. Δεν θέλουμε στη συμφωνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου να υπάρχει κάτι για την απόσπαση εργαζομένων, το οποίο να θέτει σε κίνδυνο το δικό σας το έργο και το δικό μας συλλογικό έργο για ένα νέο σύστημα ε, για το μέλλον. Αν υπάρχει στη Συμφωνία Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου, καταλαβαίνετε ότι θα είναι πιο δύσκολο μετά να αλλάξει κάτι στο μέλλον. Οπότε, εμείς πιστεύουμε ότι δεν είναι καλή ιδέα να αποτελέσει μέρος της Συμφωνίας Αποχώρησης και ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποφασιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να ληφθεί υπόψη στις μελλοντικές σχέσεις που θα έχουμε για το Ηνωμένο Βασίλειο. Γιατί είπαμε αυτό θα είναι το δεύτερο μεγάλο κεφάλαιο διαπραγματεύσεων. Το μέλλον των σχέσεών μας. Εκεί βλέπω να έχει θέση η υπόθεση αυτή. Τώρα για τους διασυνοριακούς εργαζόμενους, αυτό είναι κάτι πάνω στο οποίο πρέπει να τοποθετηθεί το Ηνωμένο Βασίλειο. Ήδη στη Συμφωνία Αποχώρησης γιατί επηρεάζει την κατάσταση πολλών ανθρώπων. Και δεν συμβαίνει αυτό τώρα προς το παρόν. Δεν έχουμε τοποθέτηση του Ηνωμένου Βασιλείου για αυτούς τους διασυνοριακούς εργαζόμενους. Και όσον αφορά το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, το είπα νομίζω και στην εισαγωγή μου, για τα δικαιώματα, τα συγκεντρωτικά, ότι η συγκέντρωση αυτή δικαιωμάτων δεν πρέπει να πληγεί εξαιτία της αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτά λοιπόν είναι τα τρία σημεία που ήθελα να ξεκαθαρίσω για να μην υπάρχει παρεξήγηση για την απόσπαση και τα λοιπά. Τώρα και κάτι για να αναφέρθηκε στο ρόλο των διαφόρων επιτροπών. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι ότι διακρίνουμε τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την αποχώρηση. Εδώ συμμετέχουν κάποιες επιτροπές πλήρως. Η Επιτροπή Απασχόλησης, η Επιτροπή ε, Πολιτικών Δικαιωμάτων ε, συμμετέχουν πλήρως και τις καλούμε στην ε, Διευθυντική Επιτροπή την κυρία Κρέσλε και τον Ζων Αρτουή που είναι οι πρόεδροι των Επιτροπών Ελέγχου Προϋπολογισμού και Προϋπολογισμών. Αυτό κάνουμε τώρα. Τώρα, όσον αφορά τις μελλοντικέ σχέσεις με τον Ηνωμένο Βασίλειο, εκεί θα εμπλακούν και άλλες επιτροπές. Αλλά προς το παρόν δεν ενθαρρύνουμε την Επιτροπή Μεταφορών, για παράδειγμα που θα μιλήσει για τον Καλάζιο Εθέρα ή την πολιτισμού που θέλει να μας πει πώς ασχοληθούμε στο μέλλον με το έρασμος κτλ. κτλ. Γιατί αυτό σημαίνει ότι έχουμε περάσει ήδη στο δεύτερο στάδιο. Μιλάμε ήδη για την μελλοντική μας σχέση. Ενώ εμείς είπαμε ότι θέλουμε να ακολουθήσουμε μια συγκεκριμένη σειρά. Ότι τώρα συζητάμε για την αποχώρηση. Και κάποιες επιτροπές συμμετέχουν πλήρως. αυτό πάει στην CCC, ε, την ε, Επιτροπή Πρόεδρων Επιτροπών, που είναι η αγαπημένη μου. Και πήγα και τους εξήγησα που βρισκόμαστε, το κάνω. Και έρχομαι και εδώ στη δικιά σας Επιτροπή και πάω και σε άλλες. Αλλά η ενημέρωση αυτή έχει να κάνει με τα συγκεκριμένα θέματα που απασχολούν τις επιμέρους επιτροπές. Δεν θέλουμε να ξεκινήσουμε εδώ όλη τη συζήτηση για, το, για παράδειγμα τι εμπορικέ σχέσει θα μπορούσαμε να έχουμε με το Ηνωμένο Βασίλειο και να αρχίσουμε συζήτηση γι' αυτό. Όχι, δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Τώρα είμαστε στη συμφωνία αποχώρησης ο κύριος Μπαρνιέ και το Συμβούλιο, μια που συμπίπτει η άποψη των τριών θεσμικών οργάνων για μια φορά, ξέρετε ότι δεν συμβαίνει αυτό πολύ συχνά, οπότε πρέπει να προχωρήσουμε με τη σειρά που έχουμε αποφασίσει. Πρώτα αποχώρηση και αν έχουμε προχωρήσει αρκετά όσον αφορά την αποχώρηση. Δεν χρειάζεται να έχει ολοκληρωθεί αυτό το κεφάλαιο, αλλά τουλάχιστον έχει προχωρήσει αρκετά. Τότε μόνο να περάσουμε στο επόμενο στάδιο που έχει να κάνει με τις μελλοντικέ μας ε, σχέσεις. Και τότε θα ρωτήσω τις διάφορες επιτροπές ποια είναι η άποψή σας, για παράδειγμα, για το Εράσμους, για τις μεταφορές, για το Blue Sky κλπ. κλπ, κλπ. Τότε θα ρωτήσω τις επιμέρους επιτροπές για την άμυνα, εξωτερικές υποθέσεις, όταν φτάσουμε στο δεύτερο σκέλος που θα είναι οι μελλοντικέ μας σχέσεις. Δεν θέλω, έρχονται κάθε τόσο οι πρόεδροι των επιτροπών και μου λένε πότε θα σας δούμε, μα δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί για να με δείτε. Τώρα έχουμε να κάνουμε με τα δικαιώματα των ε, πολιτών, τα οικονομικά, τα ελλανδικά ε, σύνορα και διάφορα άλλα ζητήματα όπως σας είπανε ναι, ο κύριος Μπούζεκ της Ήτρε Δυσκολήθηκε από μένα στην ε, Διευθυντική Επιτροπή για να μιλήσουμε για την Euratom. Γιατί αυτό είναι ένα από τα θέματα που εξετάζουμε για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Κάνω ό,τι μπορώ να και που χρειάζεται. Κύριε Μπασίρ. Είναι κρίμα που φεύγετε, εγκαταλείπετε τα κοινωνικά δικαιώματα που αφήνεται μόνος τους όλους αυτούς τους καημένους τους εργαζόμενους στην Ευρώπη χωρίς δικαιώματα. Δεν δείχνει τότε αλληλεγγύη από την πλευρά σας η αποχώρηση αυτή απέναντι στους καημένους Ευρωπαίους εργαζόμενους, αλλά τέλος πάντων είναι μια προσωπική αντίδραση αυτή. Με τον κύριο Μαν Σάιμον, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείο, ο κύριος Ντέβις και η κυρία Μέη είναι εκείνοι που συζητούν από εκείνη την πλευρά. Εγώ συναντιέμαι με την Βρετανική κυβέρνηση, περιφερειακές αρχές, την κυβέρνηση της ε, Σκοτίας, ως συντονιστής από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου τόσο πολλούς Ιρλανδούς, να ξέρετε, όσο είδα τον τελευταίο καιρό. Ε, έχω γίνει εμπειρογνώμονας τελικά για τα θέματα Ιρλανδίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Αλλά μέσα σε αυτήν την τριάδα. που ασχολούνται με το Brexit. Μπορώ βέβαια να σας πω ότι προσπαθώ να έχω όσο γίνεται περισσότερες επαφές και με άλλους. Και αυτοί του Λονδίνου, να ξέρετε, δεν είναι πάντα πιο πολύτομοι. Για να διορθώσω λίγο αυτό που είπατε εσείς για το Λονδίνο. Εσείς μιλάτε βέβαια για τους πολιτικούς στο Λονδίνο, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, αυτή είναι η αντίδρασή μου. Και σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία αυτή που μου δώσατε να έρθω και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ Γκί. Οι διαπραγματεύσει δεν θα ολοκληρωθούν σύντομα, οπότε θα σε ξαναδούμε ξανά και ξανά στην Επιτροπή μας. Καλή επιτυχία. Um, Αγαπητοί συνάδελφοι, προτείνω να συνεχίσουμε γιατί έχουμε καθυστερήσει. Can we proceed, please? Μπορούμε να προχωρήσουμε παρακαλώ. Καθίστε. συνεχίζουμε με την παρουσίαση μιας μελέτης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την απασχόληση. Μαθητεία, πρακτική και εθελοντισμός. Μία μελέτη που ζητήθηκε από το Τμήμα Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την Επιτροπή Απασχόλησης. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Τέρενς Χόγκαρτ και τον Τζάκομο Πορτολίνο, τους συντάκτες της μελέτης. Έχετε το λόγο. Ευχαριστούμε πολύ για την ε, πρόσκληση να σας παρουσιάσουμε τα ευρήματα της μελέτης για την ε, ανάπτυξη δεξιοτήτων. Εκπροσωπούμε ένα ερευνητικό ίδρυμα, το Δήμα Μπροντολίνη, Μέδρα, τη Ρώμη. Θα μιλήσω λοιπόν εκ μέρους των ε, συναδέλφων που συνέταξαν τη μελέτη ιδιαίτερα ε, εκ μέρου του Σάιμον Μπρόκ που ήταν επικεφαλής της ομάδας. Να πω καταρχάς ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον στην ε, μαθητεία, την πρακτική και τον εθελοντισμό. Ακριβώ γιατί η μετάβαση από το σχολείο στην ε, δουλειά γίνεται ολοένα και δυσκολότερη για πολλούς. Αργεί περισσότερο, καθυστερεί και είναι πιο περίπλοκη και πολλές φορές Εργοδότε ζητούν υπαλλήλου με πείρα. Και είναι η πρώτη ερώτηση που σε ρωτά ε, κάποιο ε, που τελειώνει το σχολείο, πώ θα αποκτήσω εμπειρία. Πολλέ φορέ αποκτά εμπειρία μέσω τη μαθητεία, πρακτική και του εθελοντισμού. Και πολλές φορές η εμπειρία αυτή που ε, αποκτά κάποιο μέσω της μαθητείας ή της πρακτικής είναι ακριβώς αυτό που θέλει ο εργοδότης. Γιατί πολλές φορές αυτές οι πρακτικές ασκήσεις ε, διοργανώνονται και λαμβάνουν χώρα μέσα σε μια εταιρεία που στη συνέχεια θα προσλάβει τον ε, ασκούμενο. Η μελέτη λοιπόν που θα σας παρουσιάσω εστιάζει στην συμμετοχή, στα αποτελέσματα και στην ποιότητα και στόχο έχει να εντοπίσει τις κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι υπεύθυνοι πολιτικής έτσι ώστε να μπορέσουν επιλύοντάς τες να δώσουν θετικά αποτελέσματα στους ε, συμμετέχοντες. Νομίζω πως ε, σε γενικές γραμμές είναι θετικά τα αποτελέσματα, υπάρχουν όμως ορισμένες περιπτώσεις που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή, τις οποίες θα αναλύσω αργότερα κατά τη διάρκεια της παρουσίασης. Η έρευνα. Είναι κυρίως μια ανασκόπηση της έρευνας που έχει ήδη γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε εστιάσει σε πανευρωπαϊκές έρευνες σε όλη την επικράτεια της Ένωσης, αλλά και σε συγκεκριμένες χώρες ε, με συγκεκριμένα αποτελέσματα που μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα, λόγω των διαστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα εκεί. Μετά, συζητήσαμε με διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς και δεδομένου ότι πολλές χώρες ε, έχουν και τρέχουν τέτοια προγράμματα μαθητείας ή πρακτικής. Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις και διαφορετικά διδάγματα που μπορούμε να αντιλήσουμε από τις περιπτώσει της κάθε χώρας. Κατά την διεξαγωγή της μελέτης έπρεπε να ορίσουμε το τι ε, είναι το ενδιαφέρον για την μαθητεία, για την άσκηση, ποιος είναι ο ορισμός της μαθητείας. Δεν είναι τόσο απλό στην, ε, σε γενικέ γραμμές είναι μια εναλλακτική λύση που αφορά τον ε, χώρο εργασίας, ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, ε, αποτελεί κομμάτι της επίσημης εκπαίδευσης και κατάρτισης, στο τέλος της οποίας ο μαθητευόμενος ή ο ασκούμενος λαμβάνει ένα πιστοποιητικό, ένα παραπάνω προσώμια δεξιότητα. Σε πολλές χώρες δεν υπάρχουν τέτοια προγράμματα. Ε, και αποκτά κάποιο εμπειρία στη δουλειά. Δεν υπάρχει λοιπόν ένας ε, και μοναδικός ορισμός της ε, μαθητείας, της πρακτικής άσκησης και του εθελοντισμού επίσης. Πολλές φορές ο εθελοντισμός πάει να πει ότι κάποιος προσφέρει εθελοντικά το χρόνο του, ο οποίος κάποιες φορές οδηγεί σε αποτελέσματα, σε απόκτηση δεξιοτήτων. Όμως ο εθελοντισμός είναι μια πιο ευρύτερη έννοια. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία για τους ερευνητές είναι το επίπεδο συμμετοχής σε αυτές τις ε, μαθητείες, πρακτικές και θελοντικές ε, ασκήσεις. Προσπαθήσαμε να εκτιμήσουμε τον αριθμό των συμμετεχόντων δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο νούμερο, αλλά οι εκτιμήσεις μας κυμαίνονται ανάμεσα σε 2 και 4 εκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσπαθήσαμε επίσης να, καθορίσουμε, να ε, δούμε πώς καθορίζεται αυτό, ποια είναι τα κίνητρα για την μαθητεία, την πρακτική και τον εθελοντισμό. Ποιε είναι οι απαιτήσει τη αγορά εργασίας σχετικά με τις δεξιότητες και ποια είναι τα συστήματα χρηματοδότησης ε, στις ε, διάφορε χώρε που μπορούν να επηρεάσουν άμεσα τη συμμετοχή των νέων σε αυτά τα προγράμματα. Κοιτάξαμε λοιπόν δεδομένα όλες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εκεί προέκυψε ο αριθμός ε, των 4 μέχρι 6 εκατομμυρίων συμμετεχόντων. Υπάρχει μια ανωδική τάση τα τελευταία χρόνια. Αυτά όσον αφορά την πρακτική άσκηση. Τώρα, σε γενικέ γραμμέ, ό,τι αφορά του εθελοντέ, είμαστε γύρω στο 1,5 εκατομμύριο εθελοντών. Είναι δύσκολο να υπολογίσουμε ακριβώς ε, τον αριθμό των συμμετεχόντων, όμως βλέπουμε πως ε, υπάρχει ουσιαστική συμμετοχή. Οι συμμετέχοντες είναι αρκετοί, νέοι και τα προγράμματα αυτά τους βοηθούν να κάνουν τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην απασχόληση. Οι μαθητείες έχουν σχετικά υψηλά ποσοστά επιτυχίες. Υπάρχουν ε, υψηλά ποσοστά ολοκλήρωσης του προγράμματος μαθητείας και μετά εισόδου στην αγορά εργασίας. Αυτό δεν ε, είναι κάτι που πρέπει να μας προκαλεί έκπληξη, διότι όταν μια εταιρεία επενδύει σε ένα πρόγραμμα μαθητείας, αναμένει και αποτέλεσμα. Και εάν ένας ε, μαθητευόμενος τα πάει καλά, τότε είναι αναμενόμενο και ο εργοδότης να τον κρατήσει ως ε, εργαζόμενο έπειτα. Και φυσικά όταν έχεις επενδύσει για στο να μάθεις κάποιες δεξιότητες σε έναν άνθρωπο, είναι πολύ λογικό να θέλεις και να παραμείνει κοντά σου ως ε, υπάλληλος. Υπάρχει λοιπόν μεγάλο ποσοστό επιτυχίας, υπάρχει όμως εξίσου μεγάλο ποσοστό αποχώρησης το οποίο σε ορισμένες χώρες είναι κάπως προβληματικό. Σε αυτές ε, τις ε, χώρες γίνονται έντονες προσπάθειες για να εντοπιστούν οι αιτίες του προβλήματος, οι αιτίες που κάνουν τους ε, μαθητευόμενους να αποχωρούν από τα προγράμματα, να τα παρατάνε. Προσπαθούμε λοιπόν να δούμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ε, χωρών εκείνων, να δούμε τα επίπεδα δυσκολίας της ε, μαθητείας. Πολλές φορές παρατηρούμε ότι πολλοί μαθητευόμενοι αποχωρούν από τα προγράμματα γιατί βρίσκουν μια ευκαιρία πλήρους απασχόλησης αλλού. Ενώ η ολοκλήρωση της μαθητείας έχει αβέβαια αποτελέσματα. Σε γενικές γραμμές, σε πολλές χώρες η μαθητεία θεωρείται ένα επιτυχημένος τρόπος για να γίνει μετάβαση από την εκπαίδευση στην απασχόληση. Και σε πολλές χώρες η μαθητεία γίνεται στο χώρο εργασίας με μία ήδη υπάρχουσα εργασιακή σχέση. Ο ίδιος ο φορέας απασχόλησης δηλαδή φροντίζει για την κατάρτιση του μαθητευόμενου. Τώρα, υπάρχουν διάφορες ε, πρακτικές ασκήσεις, διάφοροι τύποι πρακτικής άσκησης. Για παράδειγμα, πολλές φορές τα πανεπιστήμια προσπαθούν οι φοιτητές τους να λάβουν κάποια πρακτική άσκηση έτσι ώστε να αποκτήσουν δεξιότητες. Ε, μετά ε, η πρακτική άσκηση οδηγεί σε μία περίοδο δοκιμαστική όπου ο ασκούμενος ε, μετά από την επιτυχή ε, εκπλήρωση της πρακτικής άσκησης μπορεί να βρει απασχόληση στην εταιρεία αυτή. Πολλές φορές κάποιος μπορεί να επιλέξει την πρακτική άσκηση για να αποκτήσει δεξιότητες. Δεν γνωρίζουμε πολλά ως προς το αν η πρακτική άσκηση οδηγεί σε μόνιμη απασχόληση. Σε γενικές γραμμές όμως, όσοι ολοκληρώνουν μία πρακτική άσκηση, αποκτούν δεξιότητες, τις εκτιμούν και θεωρούν ότι τους δίνει πρόσβαση σε περισσότερες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας. Εκτιμούν λοιπόν τα προσόντα που απέκτησαν. Τώρα, εθελοντισμό. Όπως σα είπα, ο εθελοντισμό καλύπτει μια ευρύτατη γκάμα δραστηριοτήτων και είναι και τομέα που γνωρίζουμε τα λιγότερα ε, ως προς τις δεξιότητες που αποκτά ο εθελοντή. Ο εθελοντισμό όμως δίνει τη δυνατότητα στους νέους να αναλάβουν κάποιες ευθύνες μέσω της εθελοντικής εργασίας τους. Ε, πιθανώς λοιπόν έχει μεγάλη αξία για τον εθελοντή. Και όπως είπα νωρίτερα, η γενικότερη εικόνα είναι ως επιτοπλίστων θετική, με ορισμένες προκλήσεις, τις οποίες γνωρίζουμε νομίζω λίγο πολύ, και προσπαθούμε και συλλογικά και ε, ε, ατομικά να τις επιλύσουμε. Η πρώτη μεγάλη πρόκληση είναι το να γίνει ένας διαχωρισμός ε, ανάμεσα στην ουσιαστική μαθητεία πρακτική άσκηση και στην ε, κακοπληρωμένη εργασία, φτηνή εργασία. Πάντα υπάρχει ένας κίνδυνος, ε, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις πρακτικές ασκήσεις, να μην λαμβάνει ο εργαζόμενος δεξιότητες, αλλά απλά να χρησιμοποιείται ως φτηνά εργατικά χέρια. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια αποτίμηση των ε, δεξιοτήτων που αποκτά ο ασκούμενος. Επίσης, υπάρχουν διάφορα θέματα ως προς τις ίσες ευκαιρίες. Ποιος δηλαδή είναι αυτός που παίρνει τις καλές ε, θέσεις πρακτικής, ποιος είναι αυτός που παίρνει τις ε, κακές αυτό το πρόβλημα δεν ε, απαντάται τόσο συχνά στις ε, μαθητείες, γιατί πολλές από αυτές οργανώνονται από το κράτος. Δεν μπορέσαμε λοιπόν εδώ να εντοπίσουμε συστηματικές ε, καταχρήσεις του προγράμματος της μαθητείας. Υπήρξαν βέβαια διάφορα προβλήματα ως προς το ύψος των απολαβών των μαθητευομένων. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ε, πρακτικές ασκήσεις, εδώ δεν υπάρχει ε, μεγάλος έλεγχος, δεν υπάρχει ένα αριθμιστικό πλαίσιο, δεν γνωρίζουμε ακριβώς ε, τους όρους και τις προϋποθέσεις της απασχόλησης, πρακτικής άσκησης κτλ. Γνωρίζουμε λοιπόν εδώ πολύ λιγότερα. Όμως, το γεγονός ότι θεωρούν αρκετοί ότι είναι πολύτιμη η πρακτική άσκηση μας ε, δίνει μια γενικότερη θετική εικόνα. Και σε ό,τι αφορά τον αθελοντισμό, δεν γνωρίζουμε πολλά ε, ως προς τις δεξιότητες που αποκτά κανείς μέσω του αθελοντισμού. Βλέπουμε σίγουρα ότι είναι μια ωφέλιμη κοινωνικά δραστηριότητα, πως είναι ένας τρόπος να βοηθήσουμε στη μετάβαση από την εκπαίδευση στην απασχόληση, αλλά δεν έχουμε αρκετές πληροφορίες ως προς τις δεξιότητες που αποκτά κανείς μέσω του εθελοντισμού. Και είναι ένας τομέας όπου χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες. Λοιπόν, έχουμε το ερώτημα του πώς να τονίσουμε τις θετικές επιπτώσεις ε, της μαθητείας, της πρακτικής και του εθελοντισμού. Υπάρχει ένα ποιοτικό πλαίσιο που, μέσα στο οποίο προσπαθήσαμε να κινηθούμε, όπου περιέχονται κάποιοι βασικοί κανόνες, κάποιες βασικές προϋποθέσεις έτσι ώστε μετά την ολοκλήρωση μιας μαθητείας, μιας πρακτικής άσκησης, μιας εθελοντικής εργασίας να έχει ο ασκούμενος, ο μαθητευόμενος εθελοντής ε, από τα ωφέλη. Υπάρχουν όμως πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Δηλαδή, θα έπρεπε να υπάρχει, για παράδειγμα, μια σύμβαση εργασία ανάμεσα στον εργοδότη και τον εργαζόμενο ή στον μαθητευόμενο. Θα έπρεπε ο μαθητευόμενος να πληρώνεται. Ποιο είναι το ελάχιστο ε, ποσό που θα έπρεπε να λαμβάνει. Υπάρχουν λοιπόν όλα αυτά τα αναπάντητα ερωτήματα τα οποία ε, αφορούν όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου δηλαδή λειτουργούν τέτοια προγράμματα μαθητείας ή άσκησης. Και Υπάρχει φυσικά και ένα πλαίσιο που διέπει και τον εθελοντισμό αλλά και την πρακτική άσκηση. Σε γενικές γραμμές όμως υπάρχει μια παραδοχή ότι όταν γίνεται κάποια μαθητεία παίρνεις κάποιες δεξιότητες οι οποίες πιστοποιούνται κατά κάποιον τρόπο. Φυσικά όμως όπως σας είπα παραμένει αναπάτητο το ερώτημα του πώς ε, θα πρέπει να πληρώνεται ο μαθητευόμενος και αυτό γύρει και μια πληθώρα άλλων ε, ερωτήσεων, δηλαδή εάν οι απολαβές, εάν μάλλον η μαθητεία περιορίζει την πρόσβαση στην αγορά εργασίας εργοζομένων που δεν, βρίσκουν, δεν βρίσκονται σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, που θέλουν να δουλέψουν κανονικά. Αυτά ε, ως προς ε, το πεδίο εφαρμογή. Τώρα, διάφορες προτάσεις για ανάπτυξη πολιτικής. Όπως σας είπα, Παρότι οι ορισμοί δεν είναι σαφείς, υπάρχουν κάποιες ε, προσπάθειες να δοθεί ένα πλαίσιο, ένα, ένας ορισμός δηλαδή του τι ε, είναι μία μαθητεία. Υπάρχει μία γενικότερη ανωδική τάση στο να θεωρείται η μαθητεία κάτι θετικό και από τους ε, μαθητευόμενους και από τους εργοδότες. Αυξάνεται δηλαδή η ελκυστικότητα των προγραμμάτων μαθητείας, διότι σύμφωνα με τους μαθητευόμενου έχουν την ευκαιρία να δουλέψουν μαθαίνοντα και να αποκτήσουν δεξιότητες που ε, έχουν μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Όμω, πώς μπορείς να συμπεριλάβει συγκεκριμένου εργοδότες ε, σε αυτά τα προγράμματα, Πώ μπορεί να του προσελκύσει, να διευρύνει δηλαδή τη συμμετοχή από την πλευρά των εργοδοτών ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες όπως ε, γνωρίζουμε όλοι ε, θεωρούμε πάρα πολύ πολύτιμες, τις οποίες θεωρούμε τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ιδιαίτερα ε, δύσκολο θέμα είναι τα προγράμματα και θέσεις μαθητείας σε υψηλές ποιοτικά επιχειρήσεις. Υπάρχουν λοιπόν πολλά θέματα που προκύπτουν εδώ. Πώς δω δηλαδή μπορείς να διασφαλίσεις ότι θα υπάρχει ποιοτική μαθητεία, θα υπάρχουν ποιοτικές δεξιότητες, θα, υπάρχει δηλαδή ανεβασμένος πύχης ποιοτικά των προσόντων που θα αποκτά ο μαθητευόμενος. Σε ό,τι αφορά τις ε, πρακτικές ασκήσεις τώρα, Νομίζω πως εδώ μπορούμε να βελτιώσουμε πάρα πολλά και να ρυθμίσουμε επίσης, διότι πρέπει να διασφαλίσουμε πως ε, η πρακτική άσκηση δεν είναι απλά αυτή η εργασία, αλλά θα δώσει κάτι στον ασκούμενο, θα του δώσει επαγγελματικά προσόντα και δεξιότητες. Και αυτό έχει να κάνει με αυτά που έλεγα πριν, για το πώς δηλαδή μπορεί να χρηματοδοτήσεις μία πρακτική άσκηση. Διότι εάν είναι ε, αμυστή, περιορίζεται η δυνατότητα πρόσβαση στις ε, πρακτικέ ασκήσεις για ορισμένες ομάδες ε, ασκούμενων, οι οποίοι θα επωφελούνταν διαφορετικά από ένα τέτοιο πρόγραμμα. Τους κλείνουμε δηλαδή τις πόρτες όταν η πρακτική άσκηση είναι αμυστή. Και σε ό,τι αφορά τον εθελοντισμό, θα μπορούσε δυνητικά να είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για αυτήν την μετάβαση από την εκπαίδευση στην απασχόληση. Θα μπορούσε να είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για να πιστοποιηθούν οι δεξιότητες του εθελοντή. Έτσι ώστε να ανταμυφθούν οι κόποι του και η εργασία του. Εγώ ίδιος είμαι ερευνητής, οπότε δεν θα μπορούσα να ε, κλείσω χωρίς να πω ότι πάντα χρειαζόμαστε περισσότερη έρευνα, αλλά κατόπιν τούτου να πω πως αυτά τα θέματα μας απασχολούν πάρα πολύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή την εποχή. Η αγορά εργασίας ε, στους νέους είναι πάντα γεμάτη προκλήσεις και προβλήματα. Και είναι πολύ σημαντικό να ανοίξουμε τις πόρτες για τους νέους. Να τους βοηθήσουμε να αποκτήσουν πολύ σημαντικές δεξιότητες που θα τους κάνουν ελκυστικούς τους εργοδότες και τώρα και στο μέλλον. Όλη η Ευρώπη χαρακτηρίζεται από μια πληθώρα δραστηριοτήτων σε αυτούς τους χώρους. Υπάρχει μεγάλο, ε, μεγάλος πειραματισμός και νομίζω πως εδώ μπορούμε να κάνουμε πολλά και να μάθουμε ακόμα περισσότερα. Και με την εμπειρία που θα αποκομίσουμε να βελτιώσουμε τα πλαίσια που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τώρα. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και εδώ βλέπετε ένα σύνδεσμο για να διαβάζετε, αν θέλετε, τη μελέτη και ε, τα email μας έτσι ώστε να μας κάνετε οποιαδήποτε ερώτηση θέλετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Οι πολιτικές ομάδες τώρα, οι συντονιστές παρακαλώ, για σχόλια, ερωτήσεις. Από το ΕΛΚ δεν βλέπω κανένα. Ο κύριος Πάβελ από τους Σοσιαλιστές. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση και για το έργο σας. Είναι πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία αυτά. Έχω κάποιες ερωτήσεις για την αναγνώριση των προσόντων. Είπατε ότι διαπιστώνεται πως υπάρχουν πολλοί πειραματισμοί στις χώρες μέλη, διαφορετικές προσεγγίσεις Μπορείτε να μας αναφέρετε κάποια καλά παραδείγματα. Πώς η αναγνώριση αυτή δηλαδή αντιμετωπίζεται και τι συνέχεια δίνεται είτε από τους εργοδότες είτε από τους εργοζόμενους. Δεύτερον, πέρα από την αναγνώριση, πιστεύετε ότι η πιστοποίηση θα μπορεί να βοηθήσει να βρίσκει πιο εύκολα δουλειά ο κόσμος θα τον βοηθήσει. Και για την ε, αποχώρηση των νέων από το εκπαιδευτικό σύστημα, πολλούς λόγους μπορεί να φανταστεί κανείς. Εσείς τι πιστεύετε, πιστεύετε ότι υπάρχουν αυτοί οι λόγοι ευθύ εξ αρχής και μετά αποφασίζουν να σταματήσουν την εκπαίδευση ή επειδή η πληρωμή είναι πολύ χαμηλή ή δεν υπάρχει ή βρίσκουν κάποια άλλη ευκαιρία για απασχόληση και φεύγουν από αυτήν την ε, άσκηση. Υπάρχει δυνατότητα να μιλήσουμε για τις ανάγκες. Γιατί να μην τους στρέψουμε σε άσκηση, μαθητεία, πρακτική και εθελοντισμό. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας, λέει η κυρία Λαμπάτζοβα. Θα κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Κάποιες από αυτές είναι φιλοσοφικές. Μου λείπουν συγκεκριμένα παραδείγματα. Μου λείπουν συγκεκριμένα προγράμματα, σχέδια, τα οποία να λειτουργούν. Ας είμαστε ειλικρινείς, πρέπει να δούμε κάτι συγκεκριμένο. Και ακόμα, αν πούμε απλώς ποια είναι η βέλτιστη πρακτική, η καλύτερη πρακτική τέλος πάντων στις χώρες μέλη, ας το πούμε. Ας δούμε κάτι πιο συγκεκριμένο. Στην έρευνά σας ε, είδατε εσείς κάποια τέτοια καλά παραδείγματα. Καλό θα ήταν να μας το πείτε. Για μένα τώρα το μεγάλο ερωτηματικό, και εδώ είναι που περνώ πιο πολύ σε φιλοσοφικές ε, έτσι, παρατηρήσεις, δεν θέλω να μιλήσω επί πολιτικής, γιατί πολιτικά ξέρω ότι δεν θα συμφωνήσουμε. Αλλά φιλοσοφικά, η μαθητεία, η πρακτική πληρώνονται ή όχι. Αν συμφωνήσουμε ότι η μαθητεία και η πρακτική είναι κάτι χρήσιμο για να βρουν δουλειά οι νέοι και είναι κάτι αναγκαίο για να αποτελέσει μια μεταβατική περίοδο ανάμεσα στο σχολείο και την επαγγελματική ζωή, θα μπορούσα να συμφωνήσω να μην πληρώνονται. Θα τους πλήρωνε ίσως ε, το, τις δαπάνες τους, αλλά δεν βλέπω γιατί να αμείβονται, εφόσον μαθαίνουν από αυτή τη διαδικασία. Και δύο πράγματα θέλω να σας ρωτήσω. Εσείς κάνατε κάποιες συνεντεύξεις. Είπατε με τους ενδιαφερόμενους, κάνατε και με τους νέους. Απαντούν διαφορετικά οι νέοι για το θέμα της πληρωμής ή όχι της μαθητείας ή της πρακτικής. Έχετε τίποτα συμπεράσματα από τέτοιες συνεντεύξεις. Και έπειτα έχετε διαπιστώσει να υπάρχουν καταχρήσεις στη μαθητεία και την πρακτική, γιατί μπορώ να φανταστώ ότι όταν δεν υπάρχει πληρωμή μπορεί να υπάρχει κατάχρηση. Έχετε διαπιστώσει να γίνεται κατάχρηση σε τέτοιες ε, μαθητείες ή πρακτικές. Ο σκοπός είναι να βελτιωθεί η κατάσταση των νέων προκειμένου να βρίσκουν πιο εύκολα δουλειά μετά. Οπότε αν αυτός είναι ο στόχος της μαθητής και της πρακτικής θα μπορούσε να είναι και μία αμοιβόμενη. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Σιλικιώτης από την ΚΟΕ τώρα παρακαλώ. Uh, θα μιλήσω ελληνικά στη μητρική. Εγώ με τους, ε, και να ευχαριστήσω τους ειδικού που με την έρευνα παρουσιάσαν και τα στοιχεία και ως αγαπητή συνάδελφος Μαρτίνα όλα τα θέματα είναι ε, πολιτικά. Εγώ επειδή θα μιλήσω ακριβώς ότι ω αποτέλεσμα κατά την άποψή μα τη οικονομική κρίση και των πολιτικών λιτότητα, των νοφιλεύθερων πολιτικών λιτότητα που εμεί επικρίνουμε, ε, οδηγούμαστε σταδιακά σε έναν εργασιακό μεσαίωνα κατά άποψή μας. Βλέπουμε να διαλύονται δικαιώματα, να διαλύεται το κοινωνικό κράτο. Καταστράφηκαν όμω με αυτέ τι πολιτικέ πάρα πολλέ θέσει εργασία και θέσει που επέτρεπαν ε, στου νέου να ενταχθούν στον κόσμο τη εργασία. Για μα είναι πολύ θετικό πω η έρευνα δίνει και ορισμού στην μαθητεία, την πρακτική άσκηση και τον εθελοντισμό. Ε, με ανησυχεί το γεγονό ότι λόγω έλλειψη δεδομένων η έρευνα δεν μπόρεσε να δώσει σαφή εικόνα για τι ε, τάσει αναφορικά με τι πρακτικέ ασκήσει. Είναι τα ε, ε, ε, ε, ερωτήματα που έθεσε και η συνάδελφο προηγουμένω. Η αριθμοί όμω που παρουσιάστηκαν στην έρευνα, 4 με 6 εκατομμύρια νέοι, που σύμφωνα με την έρευνα μπορεί να είναι και περισσότεροι, το χρόνο σε πρακτικές ασκήσεις μας δείχνει ένα ανησυχητικό φαινόμενο αν σκεφτεί κάποιο ότι στι πλήστε αυτών των ασκήσεων συνήθω δεν παρέχουν εργασιακά δικαιώματα στου νέου. Και πολλέ από αυτέ είναι απλήρωτε. Δεν αναφέρθηκε, σημειώθηκε δηλαδή από το ερευνητή, δεν αναφέρθηκαν τα στοιχεία, αλλά γνωρίζουμε πολύ καλά και από τι χώρε μα και από τα κράτη-μέλη ότι αυτέ οι πρακτικέ ασκήσει χρησιμοποιούνται ε, ως, ε, ε, οι, νέοι ως, φθηνά εργατικά χέρια. Επίσης, παρόλο που σύμφωνα με την έρευνα το 90% των νέων που συμμετέχουν σε πρακτικές ασκήσεις θεωρούν την άσκησή τους αυτήν πολύ βοηθητική, εν τούτης, αυτή η άσκηση δεν τους οδηγεί αυτόματα σε θέση εργασίας. Διότι δηλαδή, αυτή έχει την λογική η πρακτική άσκηση. Η μαθητεία είναι να σε βοηθά, αλλά να σου ανοίγει το δρόμο, να υπάρχουν όμω αξιοπρεπεί στι για να σε οδηγήσει ε, εκεί. Αντί είναι να πληρώνουν τα αξιοπρεπή για τη δουλειά του, να απολαμβάνουν τα δικαιώματα ενό εργαζόμενου, ε, πολλέ φορέ γίνεται το μοχλό πίεση. Σε πάρα πολλά κρατημέλη έχουμε του νέου και μάλιστα πολλοί είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου να εργάζονται με προγράμμα, σε πρακτική άσκηση δίθε με 500 ευρώ ε, το μήνα αλλά να χρησιμοποιούνται σαν φθηνή εργατική δύναμη. Ε, και ε, να είναι πίεση για του υπόλοιπου εργαζόμενου. Ο κίνδυνο που νομίζω βγαίνει και από την ίδια την είναι πω οι νέοι άνθρωποι γίνονται σε πολλέ περιπτώσει ε, προϊόν εκμετάλλευση, ιδιαίτερα όταν το κράτο μέλο, και εδώ είναι που απουσιάζουν οι πολιτικέ, δεν βάζει ένα νομοθετικό πλαίσιο ε, για τι πρακτικέ ασκή εργασία. Υπάρχουν πολλά πολλά κράτη-μέλη που αυτόν τον νομοθετικό πλαίσιο απουσιάζει. Αντίθετα, οι μαθητείε σύμφωνα με την Ρέβραν εξασφάλισαν άμεση εργοδότηση, μιλώ για το σύστημα μαθητεία, για περίπου το 70% των συμμετασχόντων. Επίση, τα συστήματα μαθητεία διασφαλίζουν τα εμποδυπόδια εργασιακά δικαιώματα, έστω και αν υπάρχουν μεγάλα ποσοστά εγκατάλειψη από του νέου στη διαδικασία ε, τη μάθηση με το σύστημα μαθητεία. Και ολοκληρώνω θέτοντα μια ερώτηση στου ε, ερευνητέ ε, ε, ε, και προ του ειδικού είναι κατά πόσον μέσα από αυτή την έρευνα και τα στοιχεία που έχουν είδαν σε κάποιον κράτος μέλος να υπάρχει σε μεγάλο βαθμό διασφαλισμένο έναν είδο πρακτική άσκηση που να διασφαλίζει τα εργασιακά δικαιώματα των νέων ε, και να ανταποκρίνεται σε κρατικού σχεδιασμού, στην ανάπτυξη ενό τομέα τη οικονομία του κράτου μέλου, αλλά το κυριότερο να οδηγεί σε ασφαλή και αξιοπρεπή θέση εργασία. Εάν υπάρχουν ε, τέτοια παραδείγματα, έστω ε, και σε κάποιον από τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Thank you. And we move... Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μαρτάν τώρα από το ΙΕΝΕΦ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε καθηγητά. Σύντομα, έχω ήδη την εντύπωση ότι ο τίτλος της έρευνας δεν είναι καλός, γιατί προσπαθούμε να μπερδέψουμε την μαθητεία, την πρακτική και τον εθελοντισμό, ενώ πρόκειται για τρία διαφορετικά πράγματα. Η μαθητεία, στα γαλλικά τουλάχιστον, έχει να κάνει με τη γνώση, ότι μεταφέρουμε γνώση σε κάποιον νέο. Ε, ποια είναι το όριο, είναι 14 ή 16, μήπως είναι υπερβολικά μικρή στα 14. Μπορούμε να μάθουμε τα ίδια στα 16, για παράδειγμα, τουλάχιστον σύμφωνα με την νομοθεσία στη Γαλλία, δεν έχει δικαίωμα ένας μαθητευόμενος να ανέβει σε ένα σκαμπό ή να σερβίρει αλκοόλ. Η μαθητεία λοιπόν απευθύνεται σε νέους, πολύ νέους, για να τους μεταφέρουμε τη γνώση. Η πρακτική όμως είναι κάτι διαφορετικό. Είναι ακριβώς η θέση στην πράξη κάποιας γνώσης και να συγκρίνουμε αυτά τα οποία μάθαμε με την πραγματικότητα στον πραγματικό κόσμο, τον οικονομικό και των επιχειρήσεων. Άρα η πρακτική απευθύνεται σε κάποιον μεγαλύτερης ηλικίας για να απαντήσω στην ε, Μαρτίνα που ρωτάει θα πληρώνονται ή θα πληρώνονται οι άνθρωποι αυτοί. Μα 14 ε, ετών, γιατί τι να το πληρώσουμε, τι για να έχει ένα λίγα λεφτά στη τσέπη. Όταν όμως έχουμε να κάνουμε με κάποιον ε, που είναι 20-25 ετών, χρειάζεται χρήματα για να ζήσει. Οπότε πρέπει να αμείβεται. Και εδώ φτάνουμε και στον εθελοντισμό. Εδώ έχουμε να κάνουμε με όλους. Μπορεί κανείς να είναι εθελοντής στα 18, αλλά και στα 35 και στα 40 και στα 45. Ο εθελοντισμός είναι, θα έλεγα, κάτι που ενδιαφέρει τον άνθρωπο για τους δικούς του λόγους ή γιατί κάποιος ψάχνεται ή γιατί ψάχνει δουλειά ή γιατί θέλει εμπειρία ή πρόκειται για κάποιον ο οποίος έχει αρκετά έσοδο, οπότε δεν χρειάζεται να εργαστεί σε αμοιβόμενη εργασία και το ρίχνει στον εθελοντισμό. Είναι εντελώ διαφορετικές οι στρατηγικές και το κοινό ε, στο οποίο απευθυνόμαστε με αυτούς τους τρεις όρους. Έπειτα, και στις χώρες διαφέρουν ε, βέβαια τα πράγματα και οι κανόνες στη Γαλλία. Υπάρχει ένα συμβόλαιο για την μαθητεία και για την πρακτική και για τον εθελοντισμό. Επίσης υπογράφει κανείς ε, χαρτιά για να μπορεί να είναι ασφαλισμένος. Λέτε ότι δυσκολεύεστε να συγκεντρώσετε στοιχεία. Από τις 27 χώρες φαντάζομαι ότι τα στοιχεία διαφέρουν, αλλά αυτό όμω που συγκρατώ εγώ από τόσα μας είπατε και σας ευχαριστώ είναι ότι επιβεβαιώνεται πως παρόλα αυτά οι μορφές αυτές, ακόμα και αν δεν είναι ίδιες και δεν έχουν να κάνουν με τον ίδιο κοινό, αν μη τι άλλο αποτελούν την πύλη εισόδου συχνά στην αγορά εργασίας. Οπότε και η μαθητεία και η πρακτική και ο θελοντισμός μπορεί να έχουν αυτό το κοινό, αλλά κατά τα άλλα δεν είναι καθόλου συγκρίσιμα πράγματα. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Θα επανέλθουμε σε εσά ε, τώρα για να αντιδράσετε και να απαντήσετε στα σχόλια και τις ερωτήσεις. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορώ να απαντήσω οριστικά σε όλες αυτές, αλλά θα προσπαθήσω. Όντως, οι βέλτιστες πρακτικές είναι δύσκολο να εντοπιστούν. Υπάρχουν πολλά και διάφορα και μπορεί κανείς να προσπαθήσει να εντοπίσει προγράμματα με βέλτιστες πρακτικές, αλλά τότε χρειάζεται μια διαφορετική μελέτη. Όμως, οι μορφές ε, διαφέρουν μεν, αλλά υπάρχουν και κάποια πρότυπα, όπως το γερμανικό, για παράδειγμα, χωρίς να σημαίνει ότι η ίδια μορφή εφαρμόζεται μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλές χώρες, γιατί οι δομέ σίγουρα διαφέρουν. Δεν πρόκειται για μοντέλα που μπορεί να αντιγράψει κανεί. κανείς. Το θέμα των βέλτιστων πρακτικών είναι ακαθόδε όντω. Και χρειάζεται επιπλέον μελέτη για να δούμε τι είναι το προτιμότερο μέσα όμως σε ένα συγκεκριμένο εθνικό πλαίσιο. Τότε μπορούμε να δώσουμε συγκεκριμένα ε, παραδείγματα και καλά. Η πιστοποίηση τώρα είναι κάτι σημαντικό. Γιατί είναι δύσκολη η αγορά εργασίας για τους νέους. Και αν υπάρξει πιστοποίηση από μαθητεία, πρακτική ή εθελοντισμό, είναι κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει. Βέβαια, όταν πρόκειται για πολύ σύντομες ε, πρακτικές ή εθελοντισμό. Πρέπει να δούμε τι θα λέει το πιστοποιητικό, τι θα είναι. Το ίδιο και για το κόστος. Είναι κάτι που σίγουρα πρέπει να μελετηθεί σε λεπτομέρειες. Το θέμα τώρα της ε, αποχώρησης, της εγκατάλειψης της πρακτικής μαθητείας γιατί εγκαταλείπουν τη μαθητεία οι νέοι. Πρόκειται για εγκυμοσύνη, για παράδειγμα. Πρόκειται για το ότι οι προδιαγραφές που απαιτούνται δεν είναι προδιαγραφές στις οποίες να μπορεί να ανταποκριθεί ο μαθητευόμενος. Πάντως, αν η μαθητεία είναι σε χαμηλά επίπεδα. Λένε μερικές φορές ότι ωραία, αν δεν χρειάζεται τίποτα, ακόμα και αν πληρωθώ ένα ευρώ την ώρα, θα το πάρω. Αν βρουν δηλαδή μια τέτοια δουλειά, καταλείπουν τη μαθητεία για να πάνε σε μια δουλειά έστω και πολύ κακοπληρωμένη. Μερικές φορές φτάνουμε στο 75-80%. Και μετά σκέφτονται ότι δεν έχουν πάρει τη σωστή απόφαση. Σίγουρα κάτι δεν πάει καλά. Τώρα σε πολλές χώρες είναι ότι δεν υπάρχουν αρκετές διαθέσιμες θέσεις για μαθητεία ή και πρακτική. Οι επιχειρήσεις παίρνουν αυτούς που θεωρούν ότι ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες τους. Οπότε πώς να αυξήσουμε την πρόσβαση σε μαθητεία και πρακτική, ώστε να μπορούν να υποφεληθούν και οι δύο πλευρές. πώς να δώσεις πρόσβαση σε πιο δύσκολες περιπτώσεις. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μία μελέτη που εξετάζει το τι ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με άλλη μελέτη θα μπορούσαμε να σας δώσουμε πιο συγκεκριμένα παραδείγματα Το θέμα τώρα της πληρωμής ή όχι των πρακτικών είναι λεπτό. Αν πληρώνονται, τότε θα υπάρξουν λιγότερες διαθέσιμες θέσεις για πρακτική. Δεν θα προσφέρονται τόσο πολλές θέσεις. Από την άλλη μεριά, αν δεν πληρώνονται, κάποιες ομάδες δεν φτάνουν να έχουν πρόσβαση στην πρακτική, κυρίως όταν πρόκειται για θέσεις σε πρωτεύουσες όπου το κατάλημα κοστίζει πολύ ακριβά και άρα δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Αλλά σας λέω, συχνά οι θέσεις αυτές είναι διαθέσιμες σε πόλεις με υψηλό κόστος διαβίωσης. Δεν θα ήταν απαραίτητο να πληρώνονται όλες οι πρακτικές. Ίσως θα πρέπει να βρεθεί ένας μηχανισμός ώστε να μπορεί ο κόσμος να έχει πρόσβαση στην πρακτική χωρίς απαραίτητα να είναι ο εργοδότης αυτός ο οποίος θα πληρώνει. Αυτό θα διευκόλυνε την κατάσταση. Πάντως γενικά στη μελέτη δεν βρήκαμε κανένα στοιχείο για ε, καταχρήσεις, όπως ρωτήσατε, για συστηματικές καταχρήσεις αν μη τι άλλο. Πάντα θα υπάρχουν μονομενες τέτοιες περιπτώσεις και στην μαθητεία αυτό συμβαίνει. Γιατί αλλού είναι καλά ανεπτυγμένο το σύστημα, αλλού λιγότερο και επίσης στην περίπτωση της πρακτικής όλα εξαρτώνται από την κάθε περίπτωση. Η έρευνά μας, χωρίς να λέω ότι δεν υπάρχουν καταχρήσεις, δεν κατέληξε στη διαπίστωση συστηματικών καταχρήσεων. Τώρα, για το τρίτο σκέλος των ερωτήσεών σας. Η οικονομική κρίση φυσικά και επηρεάζει την προσφορά τέτοιων θέσεων και η αγορά δεν τα βγάζει πέρα είπαμε ότι είναι καλό για το μέλλον. Αλλά οι επιχειρήσεις, αν διαπιστώνουν ότι στο μέλλον δεν θα χρειαστούν παραπάνω προσωπικό, περιορίζουν και την προσφορά αυτών των θέσεων. Οπότε πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να καλύπτονται ε, τα κενά στην προσφορά των εργοδοτών για τέτοιες θέσεις. Όπως σας είπα, δεν διαπιστώσαμε συστηματική κατάχρηση σε αυτές τις ε, μορφές, τη μαθητεία και την πρακτική. Εμείς δεν διαπιστώσαμε κάτι τέτοιο. Τέλος, σίγουρα πρόκειται για τρεις πολύ διαφορετικές μορφές δραστηριότητας, αλλά είναι χρήσιμο να τις βάλουμε μαζί για κάποιους λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί έχουν να κάνουν όλες με τη μετάβαση των νέων από το εκπαιδευτικό σύστημα στο επαγγελματικό. Όλες έχουν να κάνουν τον ένα με τον άλλο τρόπο με τη μετάβαση αυτή. Και οι τρεις. Προσφέρουν εμπειρία, ε, πρακτική ε, άσκηση. Έχουν αυτό το κοινό. Και βοηθούν την πρόσβαση στη συνέχεια. Και είναι εθελοντές οι άνθρωποι. Σας είπα ότι ο εθελοντισμός δεν είναι τόσο για την κτήση εμπειρία. είναι περισσότερο γιατί ακολουθείς ε, αυτό που αγαπάς. Οι άλλες δύο περιπτώσεις προσφέρουν γνώση και προσόντα. Αλλά και ο θελοντισμός, γιατί τελικά μέσα από αυτό αποκτάς και παραπάνω εμπειρία. Άρα υπάρχει συσχετισμός. Συγγνώμη αν δεν μπόρεσα να απαντήσω σε όλες σας τις ερωτήσεις πλήρως. για τη μαθητεία τα στοιχεία μας είναι αρκετά καλά. Αλλά είναι δύσκολο με τις διαφορετικές τάσεις που υπάρχουν στην Ευρώπη να έχουμε εξίσου καλά στοιχεία για τον εθελοντισμό και την πρακτική. Πάντως ελπίζω να απαντήσαμε κάπως στις ερωτήσεις σας και τις απορίες σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να ασχολείται με αυτά τα θέματα τους επόμενους μήνες, τα επόμενα χρόνια, γιατί προσπαθούμε να βρούμε τρόπους μείωσης της ανεργίας και επίσης να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσει της ε, αγοράς εργασίας, το τι ζητούν οι επιχειρήσεις. Να δούμε τι και να προβλέψουμε, αν θέλετε, τι θα χρειάζεται στο μέλλον. Έχει αλλάξει ο κόσμος τα τελευταία 20-30 χρόνια και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Θα περάσουμε τώρα στο τελευταίο σημείο αυτού του απογεύματος, την παρουσίαση δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιας ε, πράξης που τελείωσε χθες που τροποποιεί τον κανονισμό του 2015. Έχουμε την ε, κυρία Τούσοβα, η οποία θα μας παρουσιάσει τις σχετικές πληροφορίες. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι πολύ που θα παρουσιάσω την τρίτη τροποποίηση του καταξουσιοδότηση κανονισμού σύμφωνα με το άρθρο 41. Αφορά την ε, υλοποίηση της δέσμευσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι θα έχουμε έναν, προσανατο... έναν προπολογισμό που θα προσανατολίζεται στα αποτελέσματα. Καλύτερη εστίαση δηλαδή στα αποτελέσματα παρά στην διαδικασία. Επίσης θα φροντίσουμε για μια ε, ταχύ εφαρμογή και ε, εξίσου γρήγορες πληρωμές μειώνοντας ε, τα ποσοστά ασφάλματος και μειώνοντας επίσης και το διοικητικό άχθος το άρθρο 41 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου αφορά, ε, αναφέρει τα ε, καταποκοπή ποσά για την επιστροφή δαπανών από την Επιτροπή στα κράτη-μέλη. Υπάρχουν ε, πολλά θετικά για αυτό το νέο άρθρο. Καταρχάς δίνει ασφάλεια δικαίου στα κράτη-μέλη και στη σχέση ανάμεσα στην διαχειριστική αρχή, το κράτος και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα προβάλλει ένσταση για τα ποσά που θα εκρίνονται σύμφωνα με τις πράξεις κατά εξουσιοδότηση. Αυτό διότι η μεθοδολογία και η απλοποιημένη διαδικασία προσδιορισμού του κόστους έχει συζητηθεί εκτενώς ε, και διμερώς με τα κράτη-μέλη. Μετά, με αυτόν τον τρόπο θα μειώσουμε τους ελέγχους και θα περιοριστούν αυτοί μόνο στον έλεγχο των αποτελεσμάτων ε, που έχουν επιτευχθεί από τα κράτη-μέλη. Οι εθνικές αρχές των κρατών μελών θα έχουν όλη την ε, ελευθερία να αποφασίσουν πώς, ε, ποια μέθοδο θα εφαρμόσουν για τον υπολογισμό των πληρωμών. Και ένα άλλο θετικό, απλοποιημένο κόστος ε, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στις περιπτώσεις ε, δημοσίων συμβάσεων. Αυτή είναι η τρίτη τροποποίηση της πράξης κατά εξουσιοδότηση που εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2015 το κύριο τμήμα της δεν έχει αλλάξει. Ακολουθήσαμε το μοντέλο του να κρατήσουμε, του να μόνο τα παραρτήματα και στην τρίτη τροποποίηση της πράξης κατά εξουσιοδότηση βλέπετε όλες τις απλοποιημένες, τους απλοποιημένους υπολογισμούς του κόστους χωρίς να χρειάζεται να ανατρέξουμε στις προηγούμενες εκδοχές του κειμένου. Μετά υπάρχουν κάποιες, ε, κάποιοι υπολογισμοί για την Σουηδία, απλοποιημένος υπολογισμός κόστους για τη Γαλλία. Το Μάρτιο του 2016 υπήρξε νέο πρόσθετο κόστος για την Τσεχία και για το Βέλγιο. Δεύτερη τροποποίηση πέρυσι τον Οκτώβριο συμπεριέλαβε πρόσθετο κόστος ε, μονάδας για την Τσεχία και την πιθανότητα για την Ιταλία, τη Μάλτα, τη Σλοβακία, τη Γερμανία και τις ε, κάτω χώρες. Σήμε... Χθες μόλις εγκρίθηκε η τρίτη τροποποίηση, η οποία καλύπτει τροποποίηση των, ε, του μονάδας για την, του, των κλιμάκων μοναδίου κόστου για τη Σουηδία. Νέε τυποποιημένε κλίμακε ε, για αρκετές ακόμα χώρες, ένα καταποκοπήν ποσό για τις κάτω χώρες που είναι κάτι καινούργιο, καλύπτει ένα νέο, μια νέα δαπάνη και η καινοτομία στον κανονισμό είναι ότι για πρώτη φορά προτείνουμε αυτήν την ε, μέθοδο υπολογισμού για την εκπαίδευση. Και για τη Σουηδία, να μπω σε λεπτομέρειες, η τροποποίηση αυτή περιλαμβάνει όλο το κόστος λειτουργίας που προηγουμένως κάλυπτε μόνο το προσωπικό ε, και την κατάρτιση. Η Τσεχία προτείνει τρία διαφορετικούς ε, τομείς, τις διαφορετικές μονάδες κόστους που ε, στηρίζουν τις επενδύσεις και την εκπαίδευση. Η Μάλ, στη Μάλτα το μοναδίο κόστος αφορά την κατάρτιση προσωπικού στις επιχειρήσεις, είτε ε, επιτόπου είτε εξωτερικά. Στην Ιταλία τρεις ε, τομείς στον χώρο της εκπαίδευσης, ε, τρεις ε, τομείς ε, για προγράμματα μαθητείας και εκμάθησης γλωσσών και τομείς για κατάρτιση νέων και διάφορα περιφερειακά προγράμματα για θέσεις διδακτορικής μελέτης μετά στην Σλοβακία υπάρχει, υπάρχουν τομείς ε, που και πάλι αφορούν την εκπαίδευση, κόστος ε, επανακατάρτισης διδασκόντων. Στην Αυστρία και πάλι εκπαίδευση, ε, απολαβές καθηγητών στην Λιθουανία επαγγελματική κατάρτιση ε, που εξαρτάται από τη διάρκεια της κατάρτισης και από το αν η ε, κατάρτιση είναι τυπική ή άτυπη. Μετά ε, κινητικότητα, μαθητεία, πρακτικές ασκήσεις για τους νέους και Ρουμανία. Μηνιαία ποσά συνδρομής σε χαμηλόμιστους εργαζόμενους. Είναι ένα, ένα πολύ βελτιωμένο, απλοποιημένο πρόγραμμα. Καλύπτει 26 κρατη Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα της ε, Eurostat. Δεν μπορούσαμε να έχουμε αξιόπιστα δεδομένα στη, για την Δανία και την Ελλάδα. Το κόστος σε μονάδα στα παραρτήματα καλύπτει ε, ετήσιο κόστος σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης σύμφωνα με τη διεθνή ταξινόμηση των ε, ε, εκπαιδευτικών πτυχίων. Βασιζόμαστε και σε εθνικές διαδικασίες. Τα κράτη-μέλη μπορούν να ζητήσουν τα ποσά αυτά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς περαιτέρω αιτιολογήσεις μόνο με τον αριθμό των εγγεγραμμένων ε, συμμετεχόντων και οι δικαιούχοι θα αποζημιώνονται με πιο απλό τρόπο, κάτι που θα δώσει περισσότερη ευελιξία και στα ίδια τα κράτη-μέλη. Είναι πρώτη φορά που προτείνουμε τέτοια πουλούστευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θεωρούμε πως θα έχουμε την ευκαιρία να ε, χρησιμοποιήσουμε τα, τις τυποποιημένες κλίμακες κόστους και σε άλλους τομείς. Και να πω επίσης ότι ήδη υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για, την, για να γίνει αυτό ένας ε, κανονισμός κατεξουσιοδότηση να καλύψει τη Γερμανία, την Κύπρο και τη Γαλλία. Αυτή τη στιγμή 13 κράτη-μέλη καλύπτονται με αυτές τις ε, απλοποιημένες διαδικασίες. Με την ε, προσθήκη της Κύπρου θα έχουμε 14 και θεωρούμε πως αυτή η συμφωνία και αυτή η πράξη κατά εξουσιοδότηση θα είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να ε, επιτύχουμε αυτή την ε, απλουστευμένη διαδικασία, να μειωθούν οι δαπάνες, να μειωθεί το διοικητικό άχθος και από την πλευρά του κράτους και από την πλευρά των δικαιούχων. Οι εκτιμήσεις, σύμφωνα με ε, τα στοιχεία που έχουμε για τα επιχειρησιακά προγράμματα και τα δεδομένα των μελετών μας, αναμένεται να καλύψουν 6,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Και ελπίζουμε μέχρι το τέλος του έτους να προσθεθούν και άλλα τρία κράτη-μέλη στον κατάλογο και να εγκρίνουμε και μία επόμενη τροποποίηση από τη στιγμή που ε, ξεκαθαριστούν όλα τα, ε, όλες οι λεπτομέρειες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι πολλή δουλειά πριν καταλήξουμε σε μια απλοποιημένη διαδικασία, αλλά έχει ενδιαφέρον και σε οικονομικό επίπεδο, γιατί αποδεικνύει ότι η εμβάθυνση στην Ευρώπη είναι κάτι που θα ωφελήσει τα κράτη-μέλη, μονομενα κρατη κράτη-μέλη. Ε, λοιπόν, κλείνουμε την σημερινή συνάντηση. Η επόμενη συνάντησή μας θα είναι 28 Σεπτεμβρίου. Θα σας γνωστοποιήσουμε σε έφετο χρόνο την ημερήσια διάταξη.